Κύριοι συνάδελφοι και κύριε Επίτροπε, θα έρθουμε στο θέμα της ημερησίας διατάξεως που αναφέρεται στον προϋπολογισμό του 2013 και θα ήθελα πρώτα να διευκρινίσω ότι μετά από την ψηφοφορία του σημερινού πρωινού για την έκθεση του συναδέλφου Γιώραν Φέρμ για σχέδιο αποφάσεως και σχέδιο κανονισμού για τα ομόλογα έργων. Θεωρούμε ότι η σημερινή ψηφοφορία αποτελεί διαπραγματευτική εντολή της ομάδας του Κοινοβουλίου με στόχο να επιτευχθεί ενδεχομένως σε πρώτη ανάγνωση μια συμφωνία σύμφωνα με την Συμφωνία 66 και το παράδειγμα 21 του ε, Κοινοβουλίου. Όλες οι ομάδες που εκπροσωπούνται από τον εισηγητή, ε, μάλλον η ομάδα ε, συνοδεύεται από τον εισηγητή και τους κύριους εισηγητέ. Θα προχωρήσουμε στην εξέταση του σχεδίου του προϋπολογισμού του 2013 που ενέκρινε μόλις σήμερα το πρωί το ε, Συλλογικό και Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ήταν κάπως ασυνήθιση διαδικασία κύριε Επιτροπέ διότι πρόκειται και για σύμπτωση ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή το προσκεκλημένος να συμμετάσχει στην ε, συνεδρίαση της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτό είχε ως συνέπεια να μην μπορέσετε να προσέλθετε ενώπιον μας παρά μόλις σήμερα το απόγευμα και αντίθετα από ότι είχαμε καταλάβει έγινε μια πρώτη παρουσίαση στον τύπο από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και από εσά πριν να έρθετε. Βέβαια, πρωταρχικά πρέπει να ε, ενημερώνετε το Κοινοβούλιο. Κάπως λοιπόν είναι δυσαρεστημένη η Επιτροπή Προϋπολογισμών, παρόλο που ήταν παρόν ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου. Δεν θα υπάρξουν βεβαίω. επιπτώσεις. Το ουσιώδες είναι το περιεχόμενο του εγγράφου. Γνωρίζουμε όλοι ότι ο προϋπολισμός 2013 θα έχει μια όλος ιδιαίτερη σημασία και στο γενικό πλαίσιο, το επίκαιρο γενικό πλαίσιο, αλλά και διότι είναι και ο προϋπολισμός της τελευταίας χρονιάς του πολιετούς πλαισίου 2007-2013 και άρα θα αποτελέσει το έτος αναφοράς για τα επόμενα χρόνια. Έτσι λοιπόν κύριε Επίτροπε σας δίνω αμέσως τον λόγο. Ευχαριστώ Αλάν, κύριος Λεβαντόφσκι. Μια σύντομη αιτιολόγηση ίσως είναι απαραίτητη, όπως εξήγησε και ο πρόεδρος της Επιτροπής σας την προηγουμένη εβδομάδα αντιμετωπίσαμε, θα πω εντό εισαγωγικών, μια νέα χορογραφία. Χωρί να σημαίνει αυτό ότι θα αποτελέσει νέα παράδοση Ότι δηλαδή ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου προσήλθε ακριβώς την ημέρα που θα πηγαίναμε και στην Επιτροπή Προϋπολογισμών πριν να βγούμε στη συνέντευξη τύπου, 11 και 30 δηλαδή, που είχε ε, προωρηθεί αρχικά η επίσκεψή μου εδώ σε εσά στην Επιτροπή Προϋπολογισμών. Αυτό κάπως ανέτρεψε την παραδοσιακή ατζέντα αλλά βέβαια ίσως δεν είναι και τόσο λάθος, διότι είναι πραγματική η πρόκληση του 2013 από πολλές απόψεις. Και γι' αυτό η στενή συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων αποτελεί και έναν από τους όρους για να φτιαχτεί ένας έντιμος ας πω έτσι προϋπολογισμός για το 2013, ένας αξιοπρεπής προϋπολογισμός. Και βέβαια η παρουσία ενός Προέδρου αν αποτελέσει νέα παράδοση ε, μέσα στα πλαίσια της συνεδριάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορούμε να ακολουθήσουμε την ίδια διαδικασία που ακολουθείτε να ανοίγουμε πρώτα στο κοινοβούλιο και μετά να ανοίγουμε πρώτα το κοινοβούλιο και μετά τα μίντια. Αυτό μπορεί χρονικά να ρυθμιστεί. Βέβαια ε, υπάρχει παραδοσιακή διαδικασία που είναι και πολύ ορθή. Τώρα να έρθω σε αυτή την εξαιρετική πρόταση του σχέδιου του προπολογισμού για το 2013 θα χρειαστεί να σας επαναλάβω την σημασία του ε, προπολογισμού αυτού που είναι διπλή. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο ετήσιος προπολογισμό, αλλά είναι και ο τελευταίος προπολογισμό που έχει συσσωρεύσει και ένα σωρό προβλήματα και μέσα στο εξαιρετικό αυτό πλαίσιο στην Ευρώπη αλλά δεν φταίει ο προπολογισμό βέβαια για τα δημοσιονομικά προβλήματα των χωρών μελών. Άλλωστε ούτε αποτελεί τη λύση των δημοσιονομικών προβλημάτων των χωρών μελών. Έχουμε υπολογίσει ότι αν πάρουμε μονάχα τους τόκους των χρεών των χωρών μελών ανέρχονται τρεις φορές στην αξία του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Τα, μόνο οι τόκοι ανέρχονται στο τριπλάσιο του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Άρα δεν είμαστε ούτε η αιτία ούτε η λύση, ο ευρωπαϊκό προπολογισμό δηλαδή. Αυτό που έχει σημασία ωστόσο είναι να επιτευχθεί μια ισορροπία ανάμεσα στη λιτότητα και στι επενδύσει. Οι αποστολέ μα στις 8 χώρε ε, των προγραμμάτων ε, μα δείχνουν καθαρά, που είναι και χώρε με τη μεγαλύτερη ανεργία, ότι η έλλειψη πιστώσεων σημαίνει εν τέλει και έλλειψη απασχόληση και έλλειψη ευκαιριών ιδίω για τι νέε γενναίε. Σε ό,τι αφορά το ύψος των πληρωμών, αυτό είναι χαμηλότερο από το ποσό που ζήτησαν οι, ε, ε, οι Επίτροποι Χάν και Τσιόλος, που είναι αυτοί τα χαρτοφυλάκια των οποίων έχουν τις μεγαλύτερες δαπάνες. Τα συζητήσαμε αυτά με τους συναδέλφους μου σήμερα. Έτσι λοιπόν και με την αύξηση που προβλέπουμε 6,8% σύμφωνα με τους υπολογισμούς για την συνοχή και για την γεωργική πολιτική, πάλι δεν καλύπτονται όλες οι ανάγκες του 2013. Θα κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να μειώσουμε βέβαια τα διοικητικά κόστη, όπως το ξέρετε κιόλας. Τα γνωρίζετε λίγο πολύ αυτά. Φτάνουμε στο τέλος της δημοσιονομικής προοπτικής με πρόσθετες ανάγκες πληρωμών. Αλλά αυτό δεν είναι και τίποτε το ασύνηθες. Δεν είναι βέβαια καμία έκπληξη. Τα γνωρίζουν αυτά 27 πρωτεύουσε των χωρών μελών. Δεν συγκρίνουμε όγκους, συγκρίνουμε τα μερίδια του συνόλου και διαγράφεται η ίδια τάση. Μπορείτε να προχωρήσετε στην επόμενη διαφάνεια. Δεν είναι ακριβώς όμως η ίδια, διότι όπως θα δείτε οι πληρωμές στην αρχή της ε, δημοσιονομικής προοπτικής υπήρχε μια απόσταση μεταξύ υποχρεώσεων και πληρωμών ήδη από το 2007 που δείχνουν και η σύγκριση δείχνει τώρα ότι η τάση είναι ίδια, δηλαδή ε, συσσωρεύονται οι πληρωμές στο τέλος της περίοδου. Όμως εδώ σπαταλήθηκε το 2007 και 2008 με καθυστερημένες α, ε, συμφωνίες για τη δημοσιονομική προοπτική που σήμανε ότι δεν εφαρμόζονταν και επομένως χρειάστηκε να επιταχύνουμε προς το τέλος και φαίνεται καθαρά το κενό αυτό. Και πέρσι, για το 2012, η απόσταση μεταξύ υποχρεώσεων και πληρωμών ήταν τη τάξη των 18 δισεκατομμυρίων ευρώ. Εμείς προτείνουμε για του χρόνου 13, αλλά έχουμε μαζέψει ένα βουνό από μη πληρωμένε υποχρεώσει. τα λεγόμενα τα λικιντέ, πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ εντωμεταξύ αυτό, τα ρευστοποιήσιμα υπόλοιπα, Χθε, στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων με ρώτησαν πολλές αντιπροσωπείες ποια είναι η λύση για αυτά τα ρέστα λικιντέ. Και η απάντησή μου ήταν ότι είναι απλό. Σήμερα θα γίνει η δοκιμασία, σήμερα θα γίνει το τεστ που θα προτείνουμε το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2013. Βέβαια δεν είναι κανένα θαύμα, είναι όμως ένα μέρος της απάντησης θα πρέπει να πληρώσουμε τις εκκρεμείς υποχρώσεις. Αλλιώς δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα του βουνού αυτού των ε, ρευστοποιήσιμων υπολείπων. Αυτά ξαναλέω για σας πιθανόν δεν είναι τίποτα το νέο, γιατί έχουν ήδη παρουσιαστεί και τώρα με τη ειδικία για το 2013. Οι κιανές γραμμές, οι, οι, οι, οι μπλε γραμμές, οι συνεχόμενοι κιανοί για το 2011 είναι αυτή που εφαρμόστηκε. Διότι δεν μπορούμε να πληρώσουμε παραπάνω από όσα έχουμε στον προπολογισμό. Αλλά η διακεκομένη γραμμή είναι ο όγκος των αξιώσεων, θεμητών αξιώσεων από τις 27 χώρες μέλη μέσα στα πλαίσια του 2011. Και βλέπουμε ότι οι θεμητές αξιώσεις που έρχονται από, από τις 27 χώρες μέλη όχι μόνο είναι πάνω από τον ψηφισμένο προϋπολογισμό, η συνεχιζόμενη, η συνεχής μάλλον κόκκινη γραμμή, αλλά και πάνω και από το σχέδιο του προϋπολογισμού για το 2011 που είχε προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και που συχνά κατηγορείται ότι κάνει υπερβολικές προβλέψεις. Είδατε ότι εν τέλει ήταν χαμηλότερη μάλιστα η πρόβλεψή της από τις ανάγκες των 27 χωρών μελών και ήταν μάλιστα και παραπάνω και από τον ε, ψηφισμένο προπολογισμό του 2012. Ποια είναι η μεθοδολογία τούτη τη φορά που νομίζω στηρίχθηκε και από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην δήλωσή του. Δεν μπορούμε να φουσκώσουμε περισσότερο τις υποχρεώσεις. Η προσπάθεια πρέπει να γίνει να περιοριστούν οι υποχρεώσεις όσο είναι δυνατόν, έτσι ώστε να μην παράγονται περισσότερες πληρωμές ε, στο μέλλον. Δηλαδή οι σημερινές υποχρώσεις θα είναι οι πληρωμές του μέλλοντος. Αλλά ποιο είναι το επίπεδο πληρωμών μας. Μιλώ για ε, ψηφισμένες υποχρώσεις του παρελθόντος. Αυτό είναι το νόημα των πληρωμών. Είναι εγκεκριμένες ψηφισμένες υποχρώσεις του παρελθόντος. Έγινε λοιπόν η προσπάθεια να περιοριστούν οι υποχρώσεις σε επίπεδο ρεκόρ από το 2007 έως το 2011 και το 2012 αύξαιναν οι υποχρεώσεις με ανοχή του Συμβουλίου σε πολύ ταχύτερους ρυθμούς. Τώρα είναι μονάχα στο 2% και να μην ξεπεράσουμε, παραπάνω, ε, να ξεπεράσουμε το ρυθμό του πληθωρισμού που αναμένεται. Για να πληρωθούν παραπάνω από τον όγκο του προϋπολογισμού, εμείς εξετάζουμε δύο πιλωτικά ε, προγράμματα. Τα ομόλογα έργων και το risk sharing instrument καταμερισμού του κινδύνου, για να δούμε δηλαδή αν οι αγορές θα αντιδράσουν και θα μας επιτρέψουν να διευρύνουμε τη δυνατότητα πληρωμών μας σε πολλούς τομείς. Αλλά ακόμα και αν αυξήσουμε τις πληρωμές, πάλι το κενό ανάμεσα σε υποχρεώσεις και πληρωμές παραμένει πάρα πολύ μεγάλο και το βουνό, ε, ίσως, ε, το κενό μάλλον, ίσως μειώνεται, αλλά εξακολουθούμε να έχουμε το πολύ μεγάλο πρόβλημα των υποχρεώσεων Γι' αυτό οποιαδήποτε προχρηματοδότηση, προπληρωμές για διάφορους τομείς για το 2014 και 2015 δεν θα είναι εφικτές, διότι αλλιώς θα έχουμε μια έκρηξη των ε, πληρωμών το 2014 και 2015. Αυτό είναι το κόστος του κενού ανάμεσα, των, ανάμεσα στις δύο αυτές ε, γραμμές. Να λοιπόν ο πίνακας ίσως από πιο μακριά να μην το βλέπετε τόσο καθαρά. Η κάτω-κάτω γραμμή είναι οι πιστώσεις κατά 6%, 6,8% επίσης, βλέπετε όμως και ποια ακριβώς μεγαλώνουν, δηλαδή η ανταγωνιστικότητα 17,8% και η συνοχή 11,7%. Αυτοί είναι οι τομείς πληρωμών που μεγαλώνουν, που αυξάνονται. Το άλλο που είναι σημαντικό για επικοινωνιακούς λόγους, αλλά και για τη σύνταξη προϋπολογισμών στο εθνικό επίπεδο, αυτά μου φαίνεται λίγο ακραία σπόρε σε περιπτώσει, αλλά ακόμα πιο δύσκολα είναι το πλασάρισμα του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, διότι η ΕΕ Ευρώπη έχει φύγει πλέον από τη μόδα και είναι ακόμα πιο δύσκολο να περάσει κανείς επικοινωνιακά τον προπολογισμό από ότι να τον συντάξει. Παρόλο λοιπόν την αύξηση των πληρωμών για το 2013, είμαστε 6 δισεκατομμύρια και παραπάνω κάτω από το όριο των δαπανών που είχε εγκριθεί το 2005 και έχουμε δηλαδή ένα περιθώριο ακόμα παρόλη αυτή την ε, αύξηση. Εδώ λοιπόν βλέπετε τι συμβαίνει και για την ανταγωνιστικότητα και για την συνοχή. Αυτός είναι και ο στόχος. Εκεί στοχεύουμε για το 2013. Κατά τα άλλα περιορίζουμε όσο αυτό είναι δυνατό. Να εδώ ο πίνακας, νομίζω τον έχετε ήδη αυτόν, δεν χρειάζεται λοιπόν να πω πολλά εδώ ότι αυξάνονται τα προγράμματα της ΚΑΠ, η διαβίου κατάρτιση επίσης αυξάνεται σημαντικά αυτή είναι η τομή όπου σημειώνονται πραγματικά μεγάλες αυξήσεις. Εδώ, όπως πρέπει να εμφανίζεται και σε κάθε παρουσίαση προϋπολογισμού, είναι η πίτα με τα κομμάτια, αλλά το έχετε και αυτό, έτσι μπορώ να συντομεύσω. Και τώρα πάμε στους τίτλους, στα heading και ίσως μπορούμε να προχωρήσουμε γρηγορότερα. Αυτά θα μελετηθούν αργότερα σε βάθος. Εδώ έχετε τον τίτλο 1α που αυξάνει σε συνολικό όγκο ετησίως, αλλά αυτό έχει εγκριθεί ήδη το 2005, έχει συμφωνηθεί το 2005 ή 6. Είχε συμφωνηθεί με το Κοινοβούλιο. Πρόκειται κυρίως για το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο, αλλά και για άλλα προγράμματα που βρίσκω ότι είναι πραγματικά κρίσιμα για την ανάπτυξη και για τις ε, δουλειές, την απασχόληση δηλαδή. Εδώ λίγο τι σημαίνει σε πρακτικούς όρους το να απευθυνθούμε σε πολλούς ανθρώπους, σε ε, πολλές κατηγορίες ανθρώπων δηλαδή, για τη συνοχή. Επίσης εδώ αυξάνεται ο όγκος μέσα στον χρόνο, πρόκειται για τις πληρωμές, αλλά αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, European Social Fund, με προσφορά σε αυτούς που είναι οι πιο ευάλωτοι. Τώρα ο τίτλος 2 και εξέλιξη μέσα στο χρόνο, όπου όμως αυτός ο τίτλος 2 δεν αποτελεί συγκέντρωση προσπαθειών αυτή τη φορά. Πρόκειται για την ανταγωνιστικότητα και τη συνοχή κυρίως. θα πρέπει να αναμένουμε και κάποιες ελλείψεις, κυρίως για την έρευνα. Γιατί πληρώνουμε ακόμα από του λογαριασμού του 2011. Ξαναπληρώνουμε τους λογαριασμούς του 2011. Και αρχίζουμε να πληρώνουμε και λογαριασμούς του 2012. και αυτό θα μελετηθεί, άρα τα περαιτέρω σχόλια ίσως δεν είναι απαραίτητα. Υπάρχουν ορισμένε εξελίξεις που θα ε, πρέπει να λάβουμε υπόψη, δηλαδή ένταξη της Κροατίας για τις υποχρεώσεις για την προενταξιακή ενίσχυση, αλλά και για τις πληρωμές. Αυτό είναι το ποσό το οποίο πραγματικά χρειάζεται ακόμα για την Κροατία και για υποχρεώσεις από την κατηγορία αυτή. Η Σερβία τώρα καταναλώνει πολλά από αυτά τα ε, προενταξιακά κεφάλαια. Μπορούμε να προχωρήσουμε τώρα στην διοίκηση. Εδώ βλέπετε ανάλυση του τι είναι κομισιόν. Επίσης τα άλλα θεσμικά όργανα περιλαμβανομένου του Κοινοβουλίου, του Κοινοβουλίου για το κόστος και ποια είναι κοινά στοιχεία. Υπάρχουν δύο κατηγορίες, τα ευρωπαϊκά σχολεία και οι συντάξεις που είναι κοινά. Και έχουμε και πιο λεπτομερή ανάλυση των δύο αυτών κατηγοριών του Κοινοβουλίου, αλλά και των άλλων θεσμικών οργάνων, στην διαφάνεια πάντα αυτή. Εδώ βλέπετε τον πίνακα που δείχνει τις προσπάθειες που κάνουμε να περιορίσουμε το κόστος, το, το διοικητικό κόστος. Όπως θα είδατε, δεν είμαι βέβαιος ότι πρέπει να αναφέρω τις περιπτώσεις, αλλά σε δύο περιπτώσεις όπου δεν υπήρχε αιτιολόγηση για αυξήσεις άνω του 1,9% του πληθωρισμού, η απόφαση που λάβαμε ήταν να κόψουμε τις φιλοδοξίες αυτών των α, θεσμικών οργάνων που ζήτησαν παραπάνω στο 1,9%. Πρόκειται για μια πραγματικά πρωτότυπη ε, ε, ενέργεια εφόσον δεν είναι αιτιολογημένες, δεν είναι δικαιολογημένες μάλλον οι δαπάνες αυτές θα πρέπει να περιοριστούμε μόνο στο ύψος του ρυθμού του, προϋπο... του πληθωρισμού. Τώρα, 12 είναι οι δικαστές βέβαια για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο που έχουν εγκριθεί. Αυτή λοιπόν είναι μια περίπτωση που γίνεται ανεκτή του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και Επίσης υψηλό κόστος μισθωμάτων, αλλά αυτό έχει σχέση με την, ε, με την ε, υπηρεσία εξωτερικών δράσεων και με την ε, καθίδρυσή της κτλ. Όμως το άρθρο 314 για πρώτη φορά χρησιμοποιείται για μια προς τα κάτω αναθεώρηση των φιλοδοξιών ορισμένων θεσμικών οργάνων. Το Κοινοβούλιο βέβαια συμμορφώνεται απόλυτα τέλεια με την από κοινού αναλυφθεί υποχρέωση και δέσμευση περισσότερο να μην ε, ζητήσουμε παραπάνω αυξήσει από τον πληθωρισμό. Τώρα εδώ για τα οργανογράμματα τώρα και όχι για τα χρήματα. Βλέπετε την προσπάθεια που κάνει η Κομισιόν ε, στην στήλη παριθμών 3. Εμείς είχαμε υποσχεθεί να μειώσουμε κατά 1% δηλαδή 263 θέσεις. Ακόμα και με τις προσλήψεις προσωπικού για την Κροατία και για το 2014 βέβαια θα προσλάβουμε, παρόλα αυτά παραμένουμε στο μείον και εξισορροπούμε κάπως άλλα θεσμικά όργανα που αυξάνουν το οργανόγραμμά τους. Το Κοινοβούλιο πάλι εδώ ευθυγραμμίστηκε απολύως απολύτως με ε, την, την αύξηση μέσα στα πλαίσια του ποσοστού του πληθωρισμού. Λαμβάνει κάποιες παραπάνω θέσεις. Βεβαίως γνωρίζω ότι η ένταξη κουρατίας θα σημάνει πρόβλημα για, ορισμένες, ορισμένα θεσμικά όργανα. Καταλήξαμε πάντως στο καθαρό αποτέλεσμα του μείον 6%. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική ανακοίνωση αυτή που σας κάνω τώρα, διότι από το 1957 η θεσμική Ευρώπη, τα όργανα της δηλαδή, διαρκώς αυξάνουν για πρώτη φορά, για πρώτη φορά στην ιστορία, από την αρχή δηλαδή της ιδρύσεως, προβλέπουμε λιγότερη απασχόληση για τον επόμενο χρόνο από ό,τι τον προηγούμενο. Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ. Εγώ το βλέπω σαν κάτι τι το αναπόφευκτο. Ούτε μπορεί να θεωρηθεί ως φετίχ η διοικητική δαπάνη. 95% ο προπολογισμό πρέπει να κατευθύνεται στι ανάγκε τη Ευρώπη και όχι των Βρυξελών και του Στρασβούργου. Χρειάζεται λοιπόν σημαντική προσπάθεια λόγω των ευαισθησιών του τομέα, της κατηγορίας αυτής. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε πώς ε, θα αντιμετωπίσουμε τα διοικητικά έξοδα εκτός ε, της κεφαλίδας 5, δηλαδή στα προγράμματα των διαφόρων κατηγοριών και βλέπετε ότι τα ερευνητικά κέντρα είχαν προτιμησιακή θέση, αλλά νομίζω ότι κάτι τέτοιο δεν θα το δεχόταν εύκολα η Utah σε σχέση με, τις αποκεντρωμένες, με τα αποκεντρωμένα ερευνητικά κέντρα έχουμε ένα μικρό μείον. Εδώ υπάρχουν θέματα που δημιουργούν αρκετές διχογνωμίες. Ως προς τη θέση 1α για το Κοινοβούλιο, το Κοινοβούλιο έχει εκφράσει το ενδιαφέρον του γιατί μιλάμε για έρευνα καινοτομία και ανταγωνιστικότητα. Όμως υπάρχουν ορισμένα προγράμματα τα οποία δεν είναι τόσο αποτελεσματικά και θα μπορούσαμε να εξοικονομήσουμε ως προς το κόστος διαχείρισης αυτών των προγραμμάτων. Αυτό αφορά και το ίτερ. Πώς μπορεί να χρηματοδοτηθεί. Θα πρέπει να δώσουμε μεγάλη μάχη για να δούμε πώς θα φτάσουμε στην καλύτερη επιλογή για το ίτερ. Σας είχα υποσχεθεί να ε, βασιστούμε σε αξιόπιστα αριθμητικά στοιχεία. Όταν μιλάμε για εξοικονόμηση απόδοσης μέσα στα πλαίσια του 7ου προγράμματος πλαισίου, εκτός και εντός, βλέπουμε αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η εφαρμογή και δυστυχώς ε, υπάρχει χαμηλή απόδοση, χαμηλότερη από την ε, προσμενόμενη. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε κατά πόσο μπορούμε να μιλάμε για 360 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή είναι η πρόταση. Φαντάζομαι τις αντιδράσεις σας αλλά θα πρέπει να προχωρήσουμε με βάση μια συγκεκριμένη πρόταση. Και να δούμε τι περιθώρια έχουμε. Εδώ έχετε πιο λεπτομεριακά στοιχεία, ε, πίνακες με βάση τον χρηματοοικονομικό προγραμματισμό. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά γνωρίζουμε ότι στο πολιετές αυτό πλαίσιο, ότι για πολλά προγράμματα το 13 θα πρέπει να κινηθούμε διαφορετικά, διότι υπάρχει χαμηλότερη απόδοση και αν θέλουμε να περιορίσουμε τις δαπάνες, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται στον ερευνητικό τομέα για ενδυνάμει εξοικονομήσεις και βεβαίως η, η διεύρυνση με την Κροατία προς την Κροατία είναι ένα θέμα που μας απασχολεί. τα στοιχεία, τα αριθμητικά στοιχεία για την Κροατία βρίσκονται στο προσχέδιο προϋπολογισμού για τα διοικητικά έξοδα, διότι οι προσλήψεις θα πρέπει να αρχίσουν από την αρχή του επόμενου έτους. Όπως, όσον αφορά τα επιχειρησιακά έξοδα, θα φτάσουμε στα 687 εκατομμύρια περίπου και θα το δούμε και με τον ε, τροποποιητικό προϋπολογισμό όταν κλείσει η διαδικασία επικύρωσης. Αυτά για την Κροατία και αυτά όλα εντάσσονται στους κανόνες του παιχνιδιού. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε. Σας ευχαριστούμε και για τους πίνακες που έχετε διανύμει. Πολλοί ζητούν το λόγο. Θα αρχίσω με τον κύριο Τζοβάνι Λαβία που είναι και ο εισηγητής μας. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Λεβαντόφσκι για αυτή την παρουσίαση και επειδή μας ε, διένει με την εισήγησή του για να έχουμε όλα τα στοιχεία μπροστά μας και να μπορούμε να τα σχολιάσουμε. Δεν μπορώ παρά να τονίσω, όπως είπε και ο πρόεδρος Λαμασούρ στην αρχή των ε, συζητήσεων και στην αρχή της συνεδρίασης, δεν μπορώ παρά να τονίσω την σημασία αυτής της πορείας, της φετινής μας πορείας, διότι είχαμε τα πρώτα στοιχεία τα πρώτα δημοσιονομικά στοιχεία από τον πρόεδρο Μπαρόζο και για 10 λεπτά ασχολήθηκε με αυτό το θέμα στη συνέντευξη τύπου και στη συνέχεια με την συνέντευξη του κυρίου Λεβαντόφσκι θα κλείσουμε έναν ασύνηθη κύκλο που δεν θα θέλαμε να επαναληφθεί. Δηλαδή, πριν δοθούν τα στοιχεία στον τύπο, πριν γίνει ένα ανακοινωθέν ε, τύπου, θα ήταν σκόπιμο να παρουσιάζονται τα στοιχεία ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτή θα ήταν και η σωστή διαδικασία την οποία θα πρέπει να ακολουθήσουμε από το επόμενο έτους. Δεν είναι εύκολο να σχολιαστεί το προσχέδιο προϋπολογισμού, διότι μόλις το λάβαμε, έχουμε τα στοιχεία εδώ και λίγα λεπτά, και θα μπορούσε κανείς να είναι ανακριβής. Φέτος έχετε απλουστεύσει κάπως τη διαδικασία, διότι σήμερα το πρωί, σε 7.30, το BBC, προτρέχοντας, μας ε, μίλησε για 6,8% ως προς τις ε, πιστώσεις υποχρεώσεων. Ε, με συγχωρείτε, πιστώσεις πληρωμών. Ένα πρώτο θέμα το οποίο θα ήθελα να μας απασχολήσει και να ρωτήσω και τον Επίτροπο, αφορά τα λεχθέντα από τον πρόεδρο Μπαρόζο στη συνέντευξη τύπου. Δηλαδή σε σχέση με τις πιστώσεις πληρωμών, τα κονδύλια, οι εγγραφές δεν είναι επαρκείς ως προς τις πραγματικές ανάγκες. Μας έλεγε ο Επίτροπος ότι το 6,8% είναι χαμηλότερο, αρκετά χαμηλότερο από αυτά που ζήτησαν οι επίτροποι υπεύθυνοι για τα χαρτοφυλάκια γεωργίας και περιφερειακής πολιτικής. Οι ανάγκες είναι πολύ ψηλότερες λοιπόν και θυμάμαι ότι Είχαμε ζητήσει από τον Επίτροπο Λεβαντόφσκι παλιότερα να είναι και υπεύθυνο και ρεαλιστής. Αυτό υπάρχει και στις κατευθυντήριες γραμμές που εγκρίναμε στην Ολομέλεια. Και αυτό το έχει αναφέρει ο Επίτροπος στην πρώτη σελίδα της απάντησής του. Ε, το 6,8% ως προς την αύξηση των πιστώσεων πληρωμών είναι ένα ανεπαρκές στοιχείο. Είναι κάτι που δύσκολα μπορούμε να προβάλλουμε προς τα έξω. Αλλά όλοι γνωρίζουμε πώς κινηθήκαμε πέρσι. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα της συνδιαλλαγής πέρσι και φτάσαμε σε ένα σημείο μη επιστροφής με αύξηση των ε, δεσμεύσεων και όχι των πληρωμών. Και τα υπόλοιπα, τα ραλ, ήταν τέτοια ώστε να μην μπορούμε πλέον να συνεχίσουμε. Άρα η πρόταση αυτή του Επιτρόπου με αύξηση 6,8% των πιστώσεων πληρωμών είναι ένα πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Επίσης, είδαμε πως έχει ο επιμερισμός, η κατανομή των πιστώσεων πληρωμών, ακολουθώντας τις κατευθυντήριες γραμμές. Είπαμε ότι πρέπει να είμαστε αποφασιστικοί προς την ανάπτυξη και την απασχόληση και στην παρουσίαση στην παρουσίασή του ο Επίτροπος καταδεικνύει ότι αυξάνονται οι πιστώσεις πληρωμών στη στήλη 1α και στο 1β ως προς τα προγράμματα όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη για απασχόληση και ανάπτυξη. Και είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό. Βεβαίως για ορισμένα προγράμματα επιφυλάσσουμε τη θέση μας, θα εξετάσουμε το θέμα εις βάθος και δεν ξέρω κατά πόσο οι συνάδελφοι είναι απόλυτα ε, ικανοποιημένοι σε σχέση με τις περικοπές στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο για την χρηματοδότηση των 360 εκατομμύριων του ΊΤΕΡ. Άρα, σε σχέση με τις κοινοπραξίες έχουν γίνει περικοπές και αυτά θα τα αποτιμήσουμε με προσοχή, με μεγάλη προσοχή στη συνέχεια. Μέσα στα πλαίσια του τριμερούς διαλόγου ε, πριν από την ψηφοφορία. Θα ήθελα να πω ότι είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος με ορισμένες θέσεις του προπολογισμού, ιδιαίτερα σε σχέση με τις ΜΜΕ, διότι θεωρώ ότι με αυτές τις πιστώσεις υποχρεώσεων μπορούμε να ανταποκριθούμε και στην απασχόληση και στην ανταγωνιστικότητα και μπορούμε να δώσουμε μία έστω και περιορισμένη απάντηση ε, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί, να βγούμε δηλαδή από την κρίση. Η ομάδα εποπτείας, υπάρχει μία ομάδα εποπτείας και υπάρχει η διάθεση απορρόφησης αυτών των κονδυλίων και μέτρων με δράσεις και ειδικά προγράμματα, τα οποία αναγράφονται εδώ. Και αυτό είναι απότοκο των όσων συνέβησαν και τις προηγούμενες μέρες της διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στη, στον πίνακα, όπου έχουμε τις αντιπαραθέσεις με τον προηγούμενο προϋπολογισμό βλέπω ότι υπάρχει μία περιορισμένη αύξηση της στήλη 2 αλλά περισσότερο της στήλη 3 για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε ως προς τη μετανάστευση, τις μεταναστευτικές ροές. Βλέπω λοιπόν ότι δίνεται και μια κοινωνική διάσταση στον προπολογισμό, κάτι το οποίο ε, εκτιμώ ιδιαίτερα. Επίσης, θα ήθελα να υπάρχει μια καλύτερη κατανομή έτσι ώστε να μπορέσουμε να σχολιάσουμε και τις διοικητικές δαπάνες έτσι ώστε η πρόταση αυτή να συμβαδίζει με τα όσα είχαμε πει για όλα τα θεσμικά όργανα για τη μείωση διοικητικών δαπανών. Ως προς τις πιστώσεις υποχρεώσεων, ζητήθηκε αύξηση της τάξης του 2% για να συμβαδίσουμε με τον τιμάριθμο και έτσι ε, να ανταποκριθούμε και πολιτικά στις πολιτικές ανάγκες. Βεβαίως θα πρέπει να μειωθεί το χάσμα μεταξύ υποχρεώσεων και πληρωμών. Και αυτό θα το δούμε και στις δημοσιονομικές προοπτικές έτσι ώστε να αυξηθούν οι πληρωμές έναντι των ε, πιστώσεων υποχρεώσεων. Είμαι πεπισμένος ότι χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη για να βγούμε από την κρίση. Αυτό είναι ένα πολιτικό μήνυμα παγώματος των δεσμεύσεων των πιστώσεων υποχρεώσεων, με συγχωρείτε. Και γι' αυτό θα πρέπει το θέμα να μας απασχολήσει περαιτέρω. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για τις λεπτομέρειες που μας έδωσε που θα αποτελέσουν αντικείμενο συζητήσεων τις επόμενες ημέρες έτσι ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα την εμβέλεια της πρότασης και να μπορέσουμε και να αντιδράσουμε κατάλληλα αποστέλλοντας το Συμβούλιο και την Κομισιόν το μήνυμά μας. Σε σχέση λοιπόν με τις ε, πληρωμές, θα εποπτεύσουμε εκ του σύνεγγι στη διαδικασία έτσι ώστε σε επίπεδο συνδιαλλαγής να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Γιατί έχουν καταβληθεί προσπάθειες και θα συνεχίσουν να καταβάλλονται για τη σωστή απόδοση και χρήση των ευρωπαϊκών και βλέπουμε ότι οι πιστώσεις υποχρεώσεων δεν έχουν σωστή ανταπόκριση στις ε, πιστώσεις πληρωμών. Δεν πρέπει να ξαναζήσουμε τα όσα γνωρίσαμε στην Επιτροπή Συνδιαλλαγής κατά την προηγούμενη χρήση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον εισηγητή. Πράγματι, Αναφέρατε ότι υπάρχουν πληροφορίες που ακούστηκαν από τον τύπο σήμερα το πρωί. Ζούμε σε μια εποχή όπου με το Twitter και τα άλλα σύγχρονα μέσα είναι αδύνατο να αποφύγουμε κάτι τέτοιο, δηλαδή όταν κάτι βρίσκεται εν εξελίξη στον εγκέφαλο ενός επιτρόπου ήδη υπάρχει στο web τώρα γιατί αυτό το 6,8% αναφέρθηκε ότι αντιστοιχεί σε 100 δις ευρώ, εδώ νομίζω θα πρέπει να γίνει μια διόρθωση. Λοιπόν, ο Επίτροπος πρέπει να αποχωρήσει σε 35 λεπτά. Θα ήθελα λοιπόν να είσαστε πολύ σύντομοι στις ερωτήσεις και παρεμβάσεις σας, έτσι ώστε να έχει χρόνο για να μπορέσει να απαντήσει. Και θα δώσω κατά προτεραιότητα το λόγο στον άλλο εισηγητή και στους σκιώδεις. Θα ήθελα όμως όλοι να είσαστε σύντομοι. Εγώ δεν θα λάβω το λόγο. Ντέρεκ. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ την uh, πρόταση αυτή του προεκολογισμού την είδα μέσω της uh, συνεντεύξης τύπου του Επιτρόπου σήμερα το μεσημέρι ο επίτροπο, Πραγματικά δεν πέρασε εύκολα σε αυτή την συνέντευξη. Έγιναν πολλά επικριτικά σχόλια, τέθηκαν πολλά δύσκολα ερωτήματα για την πρόταση αυτή του προπολογισμού. Ε, πριν κάνω εγώ τα σχόλιά μου για τον προπολογισμό για τα διοικητικά, να κάνω δύο σύντομα σχόλια για το γενικό προπολογισμό. Καλωσορίζω τα επιπλέον κονδύλια που θα πάνε ε, σε τομείς όπως η ανάπτυξη και οι θέσει εργασία. Ε, και το λέω αυτό ως μέλος που έρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί το Ηνωμένο Βασίλειο πάλι βρίσκεται σε ύφεση σήμερα. Οπότε η Ουαλία, από όπου προέρχομαι εγώ, χρειάζονται όση βοήθεια μπορείτε να, μπορείτε να τους δώσετε. Χρειαζόμαστε λοιπόν έξτρα κονδύλια για την, ε, για την πολιτική συνοχή, για το πρόγραμμα πλαίσιο 7, για την περιφερειακή ανάπτυξη, ε, ώστε να ε, ωφεληθούν και οι περιφερειακές περιοχές. Ό,τι λοιπόν πάει στην ανάπτυξη, ό,τι επιπλέον κονδύλι πάει εκεί, εγώ το καλωσορίζω. Τώρα, για τα διοικητικά κονδύλια. Ε, εγώ είμαι ο εισηγητής του Κοινοβουλίου και για άλλα τμήματα του προπολογισμού. Ξέρω ότι αυτό είναι ένα μικρό κομμάτι του προπολογισμού, μόλι 5% του συνολικού προπολογισμού πάει στα διοικητικά κόστη και ήθελα να είμαι σίγουρο ότι εμεί ω Κοινοβούλιο αλλά και όλα τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα θα μπορέσουν να δείξουν ότι όντω μπορούν να εξοικονομήσουν χρήματα και μπορούν να συμβάλλουν και στο μέλλον κάνοντα τέτοιε εξοικονομήσει. Γι' αυτό λοιπόν το Κοινοβούλιο θα πρέπει από την αρχή να κρατήσει στο, σε κάτω από 0,9 την αύξηση αύξηση του προβολισμού για του χρόνου. Αυτό φέτος το έχουμε πετύχει. Ελπίζω να μπορέσουμε και, τον, και το ε, φθινόπωρο να μειώσουμε ακόμη περισσότερο αυτό το αριθμητικό στοιχείο και να το έχουμε κάτω από 0,9%. Θα ήθελα να ρωτήσω και για τα άλλα θεσμικά όργανα κάτι, γιατί είπατε ότι μειώνεται ο, το ποσό που, που ζητάτε και το εξηγήσατε ότι δεν θα πρέπει δηλαδή να υπάρξει αύξηση πάνω του 1,9%. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το δούμε γιατί εγώ θα ήθελα να το επιτύχουμε από κοινού με τα άλλα τα θεσμικά όργανα, έτσι ώστε όλοι να βρεθούμε τελικά κάτω από το 1,9%. Ε, μιλήσατε και για το προσωπικό. Ε, μόνο κάποια από τα θεσμικά όργανα έχουν ξεκινήσει να λένε ότι θα μειώσουν το προσωπικό τους στο μέλλον, οπότε πρέπει να γίνει και άλλη δουλειά σε αυτό, ίσως από εσά. Και κάτι άλλο. Είναι σημαντικό νομίζω όλα τα θεσμικά όργανα να συνεργαστούν. Είναι σημαντικό και εσεί ω θεσμικό όργανο, αλλά και εμεί ω κοινοβούλιο να, θέσω να δείξουμε το καλό παράδειγμα. Το αίτημά μου λοιπόν, η έκκλησή μου είναι να συνεργαστούμε για τι διοικητικέ δαπάνε στο μέλλον και να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερο συντονισμό μεταξύ των ε, θεσμικών οργάνων. Να δούμε δηλαδή τα θέματα των μεταφράσεων, ε, τη διερμηνία, τα, τις ανθρώπινες, τους ανθρώπινους πόρους, ε, ε, τα θέματα των ε, υπολογιστών κτλ. Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε από κοινού για το μέλλον, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ξεκονομήσουμε χρήματα από εκεί. Ε, σας κάνω έκκληση λοιπόν σήμερα να δούμε πολύ προσεκτικά τον διοικητικό προπολογισμό, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δούμε πού μπορούν να γίνουν εξοικονομήσεις από τον προπολογισμό αυτό στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφοι. Ε, presidente, señor comisario. κυρία Σε σχέση με τα στοιχεία αυτά που λάβουμε πρόκειται για μία αξιολόγηση, συνεκτική αξιολόγηση. Θεωρώ όμως ότι μπορούμε ήδη να συναγάγουμε ότι αντικατοπτρίζει την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Γιατί ότι πρόκειται για εισηγήσεις, ζωντανές εισηγήσεις, όπου τονίζουμε τους τομείς όπου γίνεται μια ειδική προσπάθεια χρηματοδότησης έτσι ώστε να έχουμε ορισμένες κεφαλίδες, να φαίνεται ότι γίνονται επενδύσεις ως προς την εκπαίδευση, τη νεότητα, την καινοτομία και ούτω καθεξής σαν να πρόκειται για ένα γενικότερο σχέδιο και με βάση τα συνολικά στοιχεία και ε, αν συγκρίνουμε με τα στοιχεία που εδόθηκαν, βλέπουμε ότι ο προγραμματισμός παραμένει ο ίδιος ε, με το 2013 γιατί στη θέση 3 και 4 βρισκόμαστε χαμηλότερα από τα ποσά που είχαν αρχικά προγραμματιστεί και μιλάμε για μία χαμηλή για αύξηση της τάξης του 2% με μείωση στη θέση 2. Δεν έχει γίνει σημαντική προσπάθεια σε κανέναν τομέα. Δηλαδή, ως προς τους τομείς που είχαμε ορίσει ως κατά προτεραιότητα τομείς, δεν καταβάλλεται ουσιαστική προσπάθεια. Κύριε Επίτροπε, θα πρέπει αυτά που είπατε να αντικατοπτρίζονται σε αυτά που βλέπουμε ενώπιόν μας, κάτι το οποίο δεν ισχύει. Ως προς τις πληρωμές, Μιλάμε για αύξηση 6,8% το οποίο ίσως φαίνεται υψηλό, θα φαίνεται σίγουρα υψηλό στο Συμβούλιο, αλλά δεν επαρκεί, δεν αρκεί. Και νομίζω ότι η Επιτροπή, ακόμα και αν δεν αρέσει το Συμβούλιο, θα πρέπει να λάβει υπόψη τις πραγματικές ανάγκες ως προς τις πληρωμές. Δεν πρόκειται για κάτι που μπορούμε να εξοραίσουμε θα πρέπει να δούμε στις πληρωμές να καταβάλλεται πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια, κάτι το οποίο δεν βλέπουμε στα αριθμητικά στοιχεία. Και δύο ερωτήσεις πολύ συγκεκριμένες. Στον ε, ε, χρηματοοικονομικό προγραμματισμό του 2013 για, μιλούσαμε για 125 εκατομμύρια ευρώ και τώρα ε, μιλάμε για διαφορά 800 εκατομμυρίων ευρώ. Θα ήθελα να ξέρω αυτή η διαφορά πού έγκυται. Επίσης, ως προς το ίτερ. Είναι κάτι που μας απασχολεί ιδιαίτερα. Εδώ έχει γίνει μια προσπάθεια για να έχουμε εξοικονομήσεις απόδοσης. Εμένα μου φαίνονται, για... μου φαίνονται περικοπές Δηλαδή κάνουμε περικοπές σε προγράμματα τα οποία θεωρούμε προγράμματα προτεραιότητας, εκτός και εάν έχουμε αλλάξει άποψη ως προς την ιεράρχηση. Πώς ε, φτάνετε σε αυτές τις εξοικονομήσεις που εγώ ορίζω ως περικοπές, γιατί είναι ένα θέμα που έχει απασχολήσει πολύ την Επιτροπή μας. Ευχαριστούμε η Συντόνια. Ε, ε. Ευχαριστώ και εσάς κύριε Πρόεδρε και τον Επίτροπο για την παρουσίαση του θέματος. Αντίθετα ωστόσο από αυτά που είπε ο συνάδελφός μου πριν από λίγο, πιστεύω ότι η αύξηση ε, πληρωμών που προτείνεται είναι ρεαλιστική. Και και από το Συμβούλιο που λέει ότι είναι υπερβολικά υψηλή. Θα έχουμε νομίζω πολλές ευκαιρίες να το συζητήσουμε το θέμα με λεπτομέρειες, γιατί τώρα κάπως μας περιορίζει ο χρόνος. Θα θέσω ορισμένα θέματα που ελπίζω να διευκρινίσουμε, όχι σήμερα απαραίτητα, αλλά στη διάρκεια της διαδικασίας του προπολογισμού. Θα ήθελα πρώτα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την γενικότερη έννοια που δίνεται, το θέμα δηλαδή, που δίνεται στον προπολογισμό του 2013, δηλαδή διασύνδεση με ανάπτυξη και δημιουργία απασχόλησης. Αυτό ενδιαφέρει τον κόσμο, αυτό ενδιαφέρει τους Ευρωπαίους να έχουν δουλειά ή αυτοί που έχουν να την κρατήσουν. Αυτή η διασύνδεση με την ανάπτυξη και την απασχόληση είναι κάτι που πρέπει ασφαλώς να μας απασχολήσει και να το ενισχύσουμε. Θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την αύξηση των πληρωμών για την ανταγωνιστικότητα και τα προγράμματα καινοτομίας. Αυτό συνδέονται και με τα όσα είπε ο συνάδελφός μου για τις μικρές και μεσές επιχειρήσεις, καθώς επίσης και τις αυξήσεις που έχουν σχέση με το πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα υπαριθμών 7 και κάτι που με ενδιαφέρει πάρα πάρα πολύ, τις αυξήσεις για την διαβίου κατάρτιση. Όλα αυτά είναι σημαντικά και καλοδεχούμενα. Νομίζω ότι πρέπει να μιλήσουμε περισσότερο για τις απαρχές της κατάστασης στις πληρωμές. Η δική μου υπόθεση είναι ότι πρόκειται για συσσωρευμένες πληρωμές από το 2011 και 2012 που βέβαια αποκορυφώνονται τώρα στην όξυνση αυτή που θα έχουμε το 2012 και το 2013. Νομίζω ότι επίσης έχουν σχέση και με τον κύκλο ζωής πολλών προγραμμάτων κάτι το, για το οποίο μιλήσατε, αλλά πρέπει να το συζητήσουμε περισσότερο. Τι είναι αυτός ο κύκλος ζωής, είναι φυσικός, φυσιολογικός κύκλος ζωής των προγραμμάτων αυτών ή είναι γραφειοκρατικός και γιατί έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση, πώς μπορούμε να την αποφύγουμε, πώς μπορούμε να ε, ενισχύσουμε τη συνεργασία με τους ε, απολύπτες, με τους ε, απολύπτες των χρηματοδοτήσεων και με τις χώρες μέλη. Βέβαια και είναι κυρίως ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των χωρών μελών βέβαια να βελτιώσουν την ε, κατάσταση. Θα ήθελα να τονίσω ότι ασφαλώς για το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο θα είναι ένα θέμα το οποίο θα θελήσει να το εξετάσει πάρα πολύ προσεκτικά. Θα αρκεστώ για την ώρα σε αυτά και θα επανέλθω όμως κατ' επανάληψη στα θέματα αυτά. Ευχαριστώ και ευχαριστώ που είστε σύντομοι, διότι ο αγαπητός Επίτροπος δεν έχει και πολύ ώρα στη διάθεσή Ο κύριος Άλβαρο εξ ονόματος των φιλελευθέρων που έχει μέχρι τώρα έχει δείξει ε, εξαιρετική διαγωγή και περιμένει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν χρειάζεται να κοιτάει κανείς την τηλεόραση του BBC, αρκούσε να διαβάσει κανείς την Daily Telegraph από μια εβδομάδα που μιλούσε ήδη για 6,8%. Το ίδιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Παρ' όλα αυτά ευχαριστώ, ευχαριστώ και για την υποβολή του εγγράφου. Θα συμφωνήσω με την Συντόνια για την αξιολόγηση βλέπουμε κάποια κίνηση να σημειώνεται και κυρίως για τους στόχους της Ευρώπης 2020 και τα θέματα εκείνα που είναι σημαντικά για μας και για μεγάλα τμήματα της πολιτικής ομάδας, δηλαδή βλέπουμε σημαντική αύξηση για την έρευνα και ανάπτυξη. Δεν έχουμε στην Ευρώπη πολλούς πόρους και κεφάλαια παρά τα κεφάλαια που έχουμε στα κεφάλια μας, ας το πω έτσι, τα μυαλά των Ευρωπαίων δηλαδή. Αν λοιπόν δοθούν παραπάνω χρήματα σε αυτά, τα προγράμματα θα έχουμε ασφαλώς ε, βελτίωση. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι λογικό να δραστηριοποιηθούμε εντονότερα στους τομείς αυτούς. Εξάλλου δεν είμαι βέβαιος τι γίνεται με τις υποχρεώσεις πληρωμών και τις ίδιες πληρωμές. Εάν οι τιμές αυτές μπορούν να διατηρηθούν στα ύψη αυτά που είναι σωστό να προσαρμοστούν οι πληρωμές στις υποχρεώσεις που οφείλουμε να σεβαστούμε και να εκπληρώσουμε. Δεν ξέρω ωστόσο αν πρέπει να αυξήσουμε τις υποχρεώσεις πληρωμών, έστω και με περιορισμένο τρόπο, να καταφέρουμε όσο είναι το δυνατόν να κλείσουμε το κενό ανάμεσα στις υποχρεώσεις και στις πληρωμές. Να κλείσει το κενό, αυτό που δηλώσατε και εσείς ότι υποτίθεστε να κάνετε. Άλλωστε εγώ τα περιθώρια θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ μεγάλα, υπερβολικά μεγάλα. Μία ερώτηση τώρα. Δεν καταλαβαίνω πολύ καλά στον τομέα της πολιτικής συνοχής το 3,3% και το 11,7% των πληρωμών που έχετε αυξήσει. Εγώ βλέπω ήδη πολλές χώρες με τις περισσότερες να έχουν σημαντικά προβλήματα για την ίδια την εκτέλεση των προγραμμάτων. Έχει νόημα λοιπόν μια περαιτέρω αύξηση ή καλύτερα να προσπαθήσουμε ε, να ε, εκπληρώσουμε τις ισορρευτήσεις υποχρεώσεις. Ας μην βάλουμε άλλωστε και εδώ λάθος κίνητρα γιατί έχουμε ακούσει και άλλα σχόλια και έχουμε ρωτήσει τα σχόλια που έχουν λάβει δηλαδή οι χώρες μέλη ποια είναι. Εάν παραπέμπουμε στην κρίση της υπερχρέωσης, τουλάχιστον οι χώρες μέλη τότε, να εφαρμόσουν την ε, διακυβέρνηση, να εφαρμόσουν και το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, να κάνουν δηλαδή τη δουλειά τους και αυτές και όχι μονάχα να αναμένουν ενισχύσεις από τον προπολογισμό. Κάτι που δεν καταλαβαίνω επίσης, τις σημαντικές δηλαδή αυξήσεις για θέματα αλληλεγγύης και μετανάστευσης. Πάλι εδώ δεν είναι δική μας υποχρέωση να αναλάβουμε τις υποχρεώσεις των χωρών μελών. Μπορούμε να συμμετάσχουμε, μπορούμε να προτείνουμε κάποιες λύσεις, αλλά αυτά μπορεί να γίνουν μέσα από κάποια προγράμματα. Γι' αυτό δεν καταλαβαίνω πολύ καλά αυτή την μεγάλη αύξηση. Ούτε θέλουμε να είναι μέτρα τα οποία απλά να απαλλάξουν τις χώρες μέλη από κάποιες ευθύνες που έχουν οι ίδιες να ασκήσουν καλύτερες και ευφιέστερες πολιτικές και στις ε, ε, και στη μετανάστευση και ούτω καθεξής. Παρ' όλα αυτά, συνοψίζοντας, θα πω ότι χαιρόμαστε για τις αυξήσεις στην ανάπτυξη και στην έρευνα και μια πρόταση που ίσως μπορεί να υλοποιηθεί στον επόμενο προϋπολογισμό. Όταν υποβάλλεται το σχέδιο προϋπολογισμού και στις ε, και για τις συζητήσεις που κάνουμε με άλλους συναδέλφους, να κάνετε και μία αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας, δηλαδή να δείξετε τα αποτελέσματα συνεργειών του προϋπολογισμού, πώς μπορεί ενδεχομένως να ε, γίνουν, πώς μπορεί δηλαδή, σε ποιο σημείο μπορούν να φτάσουν στις χώρες μέλη, χωρίς βέβαια να μπορείτε να μαντεύσετε, δεν είστε και πυθία. Η ε, κυρία Τρίπελ. Η αύξηση των υποχρεώσεων κατά 2% νομίζω ότι είναι πολύ έτσι, συντηρητική και δεν νομίζω ότι υπάρχει ούτως ή άλλως λόγος να υπάρξει καμιά ιστερική αντίδραση σε αυτό το ποσό, είναι και κάτω από τον πληθωρισμό. Βέβαια, πάντα έχουμε να αντιμετωπίσουμε ιστερικέ αντιδράσει, ειδικά για τι πληρωμέ και το 6,8. Οπότε θα πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατό να εξηγήσουμε καλά αυτό το ποσοστό. Και αυτό θα είναι κοινή απόφαση πολιτική. Ε, έχει συμβάλει και το Συμβούλιο ω προ αυτό. Γιατί είναι προ όφελο των κρατών μελών, ειδικά τώρα να μιλήσουμε για την ε, ε, μεταρρύθμιση του προπολογισμού μέσα σε έναν καιρό λιτότητας και ύφεσης. Οπότε αυτό θα πρέπει να το τονίσουμε ειδικά για τον προπολογισμό του 2013. Πρέπει να εξηγήσουμε πώς ακριβώς μπορούμε να συνδυάσουμε και τις, ε, και τις επενδύσεις αλλά και, τις, ε, και τη λιτότητα. Νομίζω ότι αυτό θα είναι ένα πολύ σημαντικό, μια πολύ σημαντική συμβολή της Κομισιόν, ειδικά ε, για να μπορέσει να προωθήσει αυτά τα μέτρα. Παρ' όλα αυτά θέλω να προσθέσω ότι μιλούμε για τον προϋπολογισμό και, το, και συμμερίζομαι η Κομισιόν έχει θέσει και τους, ε, ε, και τους στόχους του 2020 για την εκπαίδευση, για την ανταγωνιστικότητα, για την έρευνα, για την ανάπτυξη, την κοινοτομία θα πρέπει να επενδύσουμε σε πόρου και στην τεχνολογία για να έχουμε ακόμη περισσότερε θέσει εργασία. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Οι πράσινε τεχνολογίε θα πρέπει να βοηθήσουν. Είναι κινητήριο δύναμη για να δημιουργηθούν νέε θέσει εργασία. Έχω να θέσω και δύο ε, ερωτήματα. Για τη διαβίωμα μάθηση είπατε ότι μειώνονται οι υποχρεώσει και αυξάνονται οι πληρωμές. Είναι σωστό αυτό για, την, για το εργαλείο ε, συνεργασία για την ε, ανάπτυξη. Οι πληρωμέ μειώνονται και οι υποχρεώσεις αυξάνεται. Είναι, είναι σκόπιμο να γίνει αυτό. Και δεν είμαι απόλυτα σίγουρη για την ε, αν κατάλαβα καλά όλες τις α, ε, ε, διαφάνειες. Με το Life Plus τι γίνεται για, με τις πληρωμές, μειώνονται ή αυξάνονται. Και το ίδιο για τις υποχρεώσεις, τι γίνεται. Ο κύριος Άσουερθ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, υποστηρίζω τον τίτλο που έχετε βάλει στον προπολογισμό σα, επενδύσει ε, για ανάπτυξη με θέσει εργασία. Πρέπει να επικεντρωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στου τομεί που έχουν όντω ε, να προσθέσουν αξία και έχετε δίκιο. Η ανάπτυξη και η απασχόληση είναι το νούμερο ένα. Υποστηρίζουμε λοιπόν την πρότασή σα για την ανταγωνιστικότητα, για την έρευνα και την ανάπτυξη, για τη δημιουργία θέσεων εργασία και για τη βοήθεια προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και θα ήθελα να προσθέσω ότι ε, θεωρώ ότι η ενιαία αγορά που είναι το ένα εργαλείο το οποίο πάνω απ' όλα θα πρέπει να αποτελέσει το ε, βοηθητικό εργαλείο για να περάσει από την ύφεση στην ανάπτυξη η ευρωπαϊκή οικονομία και να δημιουργηθούν θέσει εργασία, δεν τα έχει καταφέρει μέσα σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον. Παρ' όλα αυτά δεν μπορούμε να δεχτούμε την πρόταση που προσθέτει στο, ε, ε στο που έχουν τα Υπουργεία Οικονομικών των ε, κρατών μελών. Μιλούμε για δύσκολους καιρούς και όταν όλοι έχουν να αντιμετωπίσουν πραγματική λιτότητα εμείς στέλνουμε το, το λαθασμένο μήνυμα στους πολίτες όταν μιλούμε για αύξηση 7% σχεδόν. Και προφανώς αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο θα γυρίσει μπούμερανγκ σε εμά και το έχουμε ξαναδεί με τις πρόσφατες εκλογές. Κύριε Επίτροπε, καταλώ την, ε, την επιχειρηματολογία σας, ε, ομολόγα έργου, ε, εργαλείο για τον κατανομή κινδύνου. Κατανοώ αυτό που λέτε, αλλά οι ψηφοφόροι δεν θα το καταλάβουν οι ψηφοφόροι κάθε εβδομάδα εμένα με ρωτούν, όπως ρωτώ κι εγώ εσάς, γιατί δεν δείχνετε ότι μπορείτε να κάνετε το ίδιο που κάνουν όλες οι επιχειρήσεις, όλες οι τοπικές αρχές, όλες οι κυβερνήσεις των κρατών μελών. Μην ζητάτε αύξηση 7% στα έσοδα. Αποδείξτε ότι προσπαθείτε να εξοικονομήσετε 7%. Γιατί πρέπει να μπορούμε να δείξουμε στο κοινό ότι είμαστε πεπισμένοι να κάνουμε ε, περικοπές σε τέτοιους καιρούς. Και ταυτόχρονα πρέπει να είμαστε ικανοί να δείξουμε στο κοινό ότι οι δαπάνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όντως προσθέτουν, ε, έχουν προσθέμενη αξία και όντως δημιουργούν καινούργιες θέσεις εργασίας και όντως οδηγούν στην ανάπτυξη. Κύριε Επίτροπε, αυτές οι προτάσεις σας δεν με πείθουν ως προς αυτό. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Ε, η Μάρτα Ανδρέασεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, δεν έχω πιστεί από την αιτιολογία που, που δώσατε για την αύξηση των πληρωμών. Μιλήσατε για καθυστερημένες ε, αξιώσεις που ήρθαν στο τέλος ε, του πολιετούς πλαισίου, δημοσιονομικού πλαισίου. Μιλήσατε για τα ραλς, για τα ρευστοποιήσιμα υπόλοιπα που αυξάνονται. τα ρευστοποιήσιμα υπόλοιπα δεν σημαίνουν κατά και νομικές υποχρεώσεις. Πολλές φορές έχουμε υποχρεώσεις που τελικά δεν οδηγούν ε, στην ε, διεξαγωγή ενός project. Οπότε μπορείτε να μας πείτε ποια από αυτά τα ραλς όντως αποτελούν υποχρέωση. Επίσης πρέπει να είσαστε προσεκτικός με τις, τελευ... με τις αξιώσεις τελευταίας στιγμής. Το 2011 μιλήσατε για 10 δισεκατομμύρια, τώρα μας λέτε 13. Ποιο είναι τελικά το σωστό αριθμητικό στοιχείο, αλλά αυτές οι αξιώσεις η τελευταία στιγμή ίσως να είναι ο τρόπος να τα κράτη-μέλη να ισοσκελίσουν τα βιβλία τους. Η κρίση δείχνει ότι στην πραγματικότητα λίγο περιθώριο υπάρχει για συγχρηματοδότηση, οπότε πραγματικά αμφιβάλλω ότι υπάρχουν αυτές οι ε, πληρωμές τελευταίας στιγμής και ότι αυτές είναι τελικά ρεαλιστικές. Μιλήσατε επίσης για το ότι δεν έχουν γίνει οι πληρωμές 10 δισεκατομμυρίων και μετά μας είπατε ότι υπάρχει 1,5 ε, δισεκατομμύριο πλεόνασμα. Είπατε ότι αυτό οφείλεται στο ότι δεν ξέρατε ποια θα ήταν τελικά τα έσοδα. Αν δείτε όμως ε, τα, ε, τις τραπεζικές ε, ε, καταστάσεις είναι ο πιο εύκολος τρόπος για να δείτε τελικά πόσο είναι τα, πόσο είναι τα έσοδα. Ο συνάδελφος μίλησε για αποτελεσματικότητα στις δαπάνες. Η κατάσταση της Ελλάδας ας πούμε που από, την, από τότε που μπήκε στην, στην Ευρωζώνη έχει λάβει 60 δις δεν δείχνει ότι υπάρχει αποδοτικότητα τελικά στις δαπάνες. Τι θα κάνετε γι' αυτό γιατί αν ελέγξετε καλύτερα πώς δαπανώνται τα κονδύλια, θα μπορούσαμε ίσως να μην έχουμε μπει σε αυτή την κρίση ή να έχουμε ήδη βγει. Γιατί χρειάζονται χρήματα περισσότερα για την ε, διαβίω μάθηση. Έχουμε πολλούς νέους που είναι απολύτως ικανοί, έχουν ε, ε, πολύ υψηλά προσόντα. για την ανταγωνιστικότητα γιατί χρειαζόμαστε περισσότερα κονδύλια ίσως να πρέπει να είμαστε λιγότερο απαιτητικοί σε ό,τι αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η βιομηχανία είναι αυτή που πρέπει να δώσει τις θέσεις εργασίας. Όχι να δοθούν περισσότερα κονδύλια για, να, για την εκπαίδευση. Αύξηση τώρα στο διοικητικό ε, προπολογισμό για τα πάντα είναι απολύτως απαράδεκτο. Εγώ δεν μπορώ να δεχτώ αυτό το 7% ούτε θα δεχόμουν καμία αύξηση οποιαδήποτε, οποιοδήποτε ύψους. Περιμένω μείωση. Και αυτό θα συνεχίσω να πιέζω να, ε, την ε, Βρετανική κυβέρνηση να κάνει. Και επίσης θέλω να πω ότι παρόλο που ε, η Ουαλία μπορεί να χρειάζεται αυτά τα χρήματα, καλό θα ήταν η, η νοτιοανατολική Βρετανία να στείλει τα χρήματα αυτά προς την Ουαλία, γιατί από το δρόμο Βρυξέλλες-Ουαλία μπορεί να χαθούν. Θα πρότεινα στον Επίτροπο να απαντήσει σε αυτό το πρώτο γύρο ερωτήσεων και εάν παραμείνει λίγος χρόνος θα έχουμε ένα δεύτερο γύρο. Θα ήθελα μόνο να κάνω ένα σχόλιο. Ο καθένας σκέφτεται ανάλογα με τις πολιτικές του θέσεις, άλλοι θέλουν περισσότερα, άλλοι λιγότερα χρήματα. Υπάρχει μία αρχή στο ρωμαϊκό δίκαιο που δεν αρνίκει, που δεν ισχύει στις χώρες ε, του εθιμικού δικαίου που λέει ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε σε μία δίκη κάποιος να κατηγορήσει κάποιον άλλον για τα δικά του τα ίδια σφάλματα. Αυτό ακριβώς κάνουν ορισμένες κυβερνήσεις. Δηλαδή έρχονται στην Επιτροπή, ζητάν χρήματα για μια περιφέρεια, για ένα ερευνητικό πρόγραμμα, για τη γεωργία και στη συνέχεια προσάπτουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δίνει θετική συνέχεια σε αυτά τα αιτήματα. Και το πολιτικό μήνυμα είναι ε, ας είστε σοβαροί, μην τιμάτε τις υποχρεώσεις σας. Είναι αυτό ακριβώς σαν να λένε ορισμένα κράτη-μέλη και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πολιτικά διλήμματα και προβλήματα. Σας ευχαριστώ για το τελευταίο σας, για όλα και για το τελευταίο σας σχόλιο, γιατί δείχνει το, καταδεικνύει το γεγονός ότι διανύουμε μια κατάσταση σχιζοφρενική ως προς τον προϋπολογισμό. Και έγινε λόγος για το ότι υπάρχουν προτιμησιακές σχέσεις με το Κοινοβούλιο εναντί του τύπου. Νομίζω όμως ότι αυτό σχετίζεται με προσωπικές προσκλήσεις προς τον πρόεδρο, αλλά φυσικά με σας πρέπει να συζητιέται καταρχήν το θέμα του προϋπολογισμού. Δεν είμαι υπεύθυνο ε, για αυτή την διαρροή που έγινε προς τον τύπο. Είναι σαν να πρόκειται, σαν για μια διαδικασία ε, δολιοφθορά. Σε πάση περιπτώσει, θυμόσαστε ότι στις προηγούμενες δημοσιονομικές προοπτικές δεν υπήρχε τέτοια διαρροή. Αυτή τη φορά δεν ξέρω, διέρευσαν κάπως τα πράγματα, βρέθηκαν ε, εκτός ελέγχου. Σε σχέση με το 6,8% που είπε ο κύριος Λαβία, βεβαίως μπορείτε να το αμφισβητήσετε. Εμείς είμαστε αισιόδοξοι και θεωρούμε ότι το 6,8% αρκεί για το 2013. Εάν δεν επαναλάβουμε την ιστορία του 2012. Δηλαδή θεωρούμε ότι με το διορθωτικό προϋπολογισμό φέτος θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε και θα γίνει αποδεκτός, όπως ισχύει στο τέλος των ε, δημοσιονομικών προοπτικών. Και η Συντόνια το ανέφερε αυτό. Και προς την κυρία Άντρισεν θα ήθελα να πω το εξής. Μιλάμε για 15 εκατομμύρια ε, ευρώ. Υπάρχουν συγκεκριμένες αξιώσεις ως προς τη συνοχή για τις τελευταίες εβδομάδες του 2011. Ως προς 10,9 δεν μπορέσαμε να καταβάλουμε τα ποσά είτε γιατί δεν υπήρξε ευελιξία, είτε επειδή δεν, υπάρχουν, δεν υπήρχαν χρήματα. Καταβάλαμε τα 5 από τα 10 εκατομμύρια το Δεκέμβριο, όπως είχαν εγγραφεί. Υπήρξαν ελλείψεις. Τώρα έχουμε ελλείψεις στην αρχή και η Συντόνια γνωρίζει πολύ καλύτερα πώς λειτουργούν τα πράγματα, πώς δηλαδή φτάνουμε σε αυτή τη διαδικασία ορίμανσης. στην αρχή. Έχουμε σωστή απορρόφηση, στο τέλος δυστυχώς υπάρχουν ελλείψεις. Αν όμως το τέλος του έτους έχετε έσοδα από κυρώσει στον ανταγωνισμό. Είχαμε 700 εκατομμύρια που συνέλεξε ο κύριος Αλμούνια. Είχαμε αυτές τις ε, χρηματικές κυρώσεις. Αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσαν να γίνουν ε, πληρωμές από αυτά τα ποσά. Έτσι αυτό αποτέλεσε πλεόνασμα. Είχαμε 400 εκατομμύρια για τις μισθολογικές προσαρμογές στα διάφορα θεσμικά όργανα. Ε, δεν μπορέσαμε να απορροφήσουμε αυτά τα ποσά, γι' αυτό θεωρήθηκε ότι υπάρχει πλεόνασμα. Ίσως αυτό να είναι και ένα θετικό μήνυμα. Εν πάση περιπτώσει, το 12 υπήρξε μεγαλύτερη εισφορά των κρατών μελών. Υπάρχει ένα ποσοστό ανελιξίας, θα μπορούσα να πω, να υπάρχει περιορισμένη απορρόφηση, περιορισμένη δαπάνη, αλλά στο τέλος να έχουμε ελλείψεις δηλαδή δεν μπορέσαμε να ανταποκριθούμε στις αξιώσεις στο τέλος του 2011. Για να είμαστε αξιόπιστοι λοιπόν θα πρέπει και όπως είπε ο έχει απόλυτο δίκιο, θα πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες, αν και πιστεύω ότι τα κράτη-μέλη, ορισμένα κράτη-μέλη έχουν ένα είδος ιδεολειψίας με αυτές τις μικρές δαπάνες, δηλαδή μιλάν για ανύπαρκτες εξοικονομήσεις δεν πρόκειται για υψηλά ποσά. Έγινε λόγος για 20 εκατομμύρια αποταμιεύσεις, αλλά δεν υπήρχαν ως προς τις διοικητικές δαπάνες. Εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να καταβληθεί αυτή η προσπάθεια. Ε, αναφερθήκαμε σε αυτό το θέμα και στην Επιτροπή Περιφερειών που ήθελε οι αυξήσεις να είναι πάνω από τον τιμάριθμο. Εμείς είπαμε ότι θα πρέπει να αρκεστούμε στον τιμάριθμο και ίσως το μέλλον θα πρέπει να μας απασχολήσει ως προς την προστασία των δεδομένων. Βρήκαμε. Λοιπόν, τις σωστές λύσεις ως προς την προστασία των ε, δεδομένων. Η Άιντερ είπε ότι δεν ανταποκριθήκαμε όπως έπρεπε. Συμφωνώ με τον κύριο ε, Άλβαρο, ο οποίος είπε ότι ποτέ δεν ήμασταν τόσο επιλεκτικοί όταν επιλέγουμε τους κερδισμένους και τους ιτημένους. Επίση, σε σχέση με το Ταμείο για τη Ζάχαρη, δεν ανταποκριθήκαμε απόλυτα και με το ίτερ θα πρέπει να δούμε πώς θα ανταποκριθούμε. Βρισκόμαστε στην απαρχή των συζητήσεων. Εν πάση περιπτώσει ήμασταν πολύ επιλεκτικοί και προσπαθούμε να μην ζημιώσουμε προγράμματα. Εάν υπάρχουν περιθώρια ελιγμών, ιδιαίτερα για, το, για διοικητικό κόστος υποστήριξης, έχει καλός. Δεν θέλουμε όμως να ζημιώσουμε τα προγράμματα της κατηγορίας 1α. Μιλάμε για 360 εκατομμύρια, αλλά θα πρέπει να ε, προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε όπως πρέπει. Μπορούμε λοιπόν να επικεντρωθούμε στο ίτερ πλέον για ένα χρόνο. Δεν έγραψα όλες τις ε, ε, ερωτήσεις σας, ε, προσπάθησα, αλλά δεν τις κατέγραψα όλες. Το Life Plus ακολουθεί ανωδική πορεία και στη Χέλγκα στον επόμενο γύρο θα απαντήσω για να σας πω πώς έχει κατανομή των δαπανών για αυτή την πρόταση. Δεν έχω πολύ χρόνο τώρα να το διερευνήσω. Αυτή τη στιγμή δηλαδή, να σας απαντήσω τώρα. Μιλάμε για έναν χρηματοδότη μηχανισμό. Ήταν σαν να πρόκειται για ένα φετίχ. Έχουμε υποχρεώσεις για το 2013 και ούτω καθεξής. Τώρα υπάρχει μία διαφοροποίηση αλλά αυτό δεν τα λέμε προς τα έξω σε σχέση με τον χρηματοοικονομικό προγραμματισμό. Δηλαδή υπάρχει ένα συσχετισμός με τον προϋπολογισμό του 2012. Και βεβαίως έχουμε και τους Βρετανούς φίλους που αναφέρθηκαν στα τέλη του 2011. Νομίζω ότι δόθηκε η απάντηση αλλά υπάρχει μια σχιζοφρενική τάση, γιατί χτες στο Λουξεμβούργο με ρωτούσαν συνέχεια τι πρέπει να κάνουμε με τα υπόλοιπα προς τα ραλ. Η κυρία Άντρισεν έχει δίκιο, δεν πρόκειται για μελλοντικές καταβολές. Το 90% οδηγεί σε μελλοντικές πληρωμές, αλλά ίσως έχουμε και υποχρεώσεις. Γι' αυτό συστέλουμε και τις μελλοντικές ε, υποχρεώσεις έτσι ώστε να μην πρόκειται για ένα πολύ επώδυνο εγχείρημα. Αλλά για να επιλύσουμε τα ραλ, τα υπόλοιπα προς εκαθάριση, πρέπει να αυξήσουμε τις πληρωμές. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Δεν βλέπω άλλη λύση σε σχέση με τους ελέγχους, με το νόμιμο, με τις αξιώσεις πληρωμών. Αυτή είναι η απάντησή μου προς τα, ως προς τα ΡΑΛ. Δεν απάντησα σε όλα τα θέματα ίσως. Αλλά επειδή είμαι, ε, μια συνάντηση με το με έναν συνάδελφο από την Ουγγαρία, με έναν υπουργό. Θα ήθελα να μην καθυστερήσω τώρα, θα πρέπει να τον συναντήσω στο Μπερλεμόν και έχω ήδη αργήσει λιγάκι. Ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα εδώ και ξεπεράσατε και το χρόνο που μπορούσατε να μείνετε. Ε, αναλαμβάνω εγώ την Προεδρία, οπότε να ακούσουμε όσους έχουν ζητήσει το λόγο. Νομίζω ότι θα έχουμε αρκετό χρόνο. Ε, και είναι σημαντικό εμείς ε, ως ε, κοινοβουλευτικοί να, είναι, να ξεκαθαρίσουμε το τι τελικά θέλουμε. Γιατί το φθινόπωρο θα βρεθούμε προ του ερωτήματος τι θέλουμε τελικά. Θέλουμε πάλι να κάνουμε αυτό που κάναμε τα τελευταία δύο χρόνια και θα πάμε μπροστά από το Συμβούλιο και θα πούμε «Αχ, ε, δεν, ε, θα, δεν μπορούμε να προσθέσουμε άλλη κρίση στην ήδη υπάρχουσα κρίση και γι' αυτό ε, πρέπει να ικανοποιήσουμε το Συμβούλιο ή θέλουμε να πούμε εμείς με το μικρό μας τον προπολογισμό μπορούμε αν όντω τον εφαρμόσουμε σωστά και τακτικά να κάνουμε πολλά καλά πράγματα. Αλλά αν το προτιμήσουμε αυτό τότε θα πρέπει να τηρήσουμε αυτή τη στάση, να την υπερασπιστούμε. Οπότε πρέπει να δούμε τι ακριβώς ε, θα γίνει. Εγώ αυτές τις δύο ε, τύπου και του πρόεδρου Μπαρόζο που ήταν μαζί με τον ε, πρόεδρο Σούλτς και την ε, συνέντευξη τύπου του Λεβαντόφσκη της είδα. Δεν θεωρώ ότι ήταν ανάγκη αυτή η πρώτη ε, συνέντευξη τύπου να γίνει, γιατί και οι δύο, και ο Σούλτς και ο Μπαρόσο, μίλησαν για το δικό μας το προπολογισμό. Ναι, αλλά όχι για το προπολογισμό του 2014, αλλά μίλησαν για αρχές. Και πώς ακριβώς εμείς αυτές τις αρχές, δηλαδή την, αν είμαστε υπέρ της, της, αύξησης του προπολογισμού ή της μείωσης αυτού, πώς πρέπει να, το, να την αξιολογήσουμε. Και εγώ πρέπει να πω ότι ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου έχει την πλήρη στήριξή μου, ο πρόεδρος της Κομισιόν είπε το ίδιο, αλλά το είπε ξεκάθαρα και ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου. Οπότε πραγματικά χαίρομαι που τον έχουμε ως πρόεδρο του Κοινοβουλίου. Jetzt noch zum Haushaltsentwurf 2013. Τώρα για τον προπολογισμό 2013. Θα δούμε. Είναι αμυντική η θέση που έχουμε λάβει. Εντάξει, δεν ακούγεται αυτό πολύ καλά για το Συμβούλιο, γιατί ούτως ή άλλως το Συμβούλιο δεν καταλαβαίνει και περί τίνος πρόκειται. Μιλούμε για αύξηση 6,3% στις πληρωμές. Προφανώς αυτό δεν ακούγεται καθόλου καλό, αλλά δεν είναι, δεν είναι έτσι. Αν δούμε για τον επόμενο χρόνο τι δημοσιονομικό πλαίσιο έχουμε ενισχύει και η Κομισιόν ταυτόχρονα μας προτείνει 2,5 δισεκατομμύρια για υποχρεώσεις και πάνω από 6 δισεκατομμύρια για πληρωμές. Ε, συγγνώμη, ας μας πει η Κομισιόν τότε πού είναι αυτό μέσα στον προπολογισμό και από πού προκύπτει και μετά μιλούμε για τους ε, τίτλους για την ε, νεολαία μας. Νομίζω λοιπόν ότι αυτός ο προπολογισμό είναι πραγματικά πάρα πολύ συντηρητικός και θα πρέπει αυτό να το υπερασπιστούμε. Να μην είμαστε μονίμως με την πλάτη στον τοίχο, να μην λέμε συνέχεια δεν εξοικονομήσαμε αρκετά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ευρωπαϊκός προπολογισμό δεν είναι για να κάνει περικοπές, επειδή καταρχάς δεν χρωστάει και επειδή είναι ο μοναδικός προπολογισμό σε όλη την Ευρώπη που μπορεί να επενδύσει. Τελεία λοιπόν. Επόμενος, ο Uh, Ευχαριστώ, ο κύριος Γκοντμάνης. Ο Επίτροπος ε, έφυγε, αλλά ξέρω ότι έχουμε εκπροσώπους της Κομισιόν εδώ, οπότε οι εμπρευνόμονες ίσως θα μπορούσαν να μου απαντήσουν. Το βασικό πρόβλημα που βρίσκω εγώ είναι τα ρευστοποιήσιμα υπόλοιπα. Πρέπει να το ξαναδούμε πολύ στενά το θέμα αυτό. Γιατί αν υπολογίσουμε μαθηματικά, έχουμε 207 τα οποία θα πάνε στην έρευνα, στην συνοχή και σε άλλα, άλλους τομείς. Κάποιοι συνάδελφοι λένε ότι αν δεν είναι νομική αυτή η υποχρέωση μπορεί και να μην πληρωθεί. Ο, Επιτροπε, ο Επιτρόπος είπε ότι είναι θεμητή η υποχρέωση. Οπότε από ό,τι καταλαβαίνω εγώ η αύξηση των πληρωμών στο 2013 μπορεί να υποστηριχθεί από το Συμβούλιο ότι, μόνο λέγοντα ότι αυτά τα, αυτά τα χρήματα θα πάνε πίσω στα κράτη-μέλη και δεν θα, πάνε, δεν θα χρησιμοποιηθούν για κοινή χρήση. Ε, σημείο 2 πρέπει να το υποστηρίξουμε. Έτσι, εγώ είμαι φιλελεύθερος, αλλά διαφωνώ με τον κύριο Άλβαρο. Έχουμε διχασμένε απόψει ε, στου φιλελεύθερου για την πολιτική συνοχή και την ε, χρηματοδότηση, αλλά εντάξει, αυτά είναι φυσιολογικά, γιατί μιλούμε για ε, όσου καταβάλουν στον προπολογισμό και όσου λαμβάνουν από τον προπολογισμό. Προφανώ είναι διαφορετικέ απόψει. Αλλά αν η Κομισιόν μα πει ότι θα υπάρξει έλλειμμα, ακόμα και με την αύξηση των πληρωμών 6,8, έλλειμμα στην εφαρμογή αυτών των, στην υλοποίηση αυτών των προοπτικών, τότε θα πρέπει να μας πει η Κομισιόν πώς αυτό σχετίζεται με το επόμενο πολιετές πλαίσιο. Γιατί αν δεν γίνουν οι πληρωμές και σύμφωνα με όλους τους ε, κανόνες, εν πλας, εν συν 2, εν συν 3 ε, και με τα χρονικά όρια επίσης που ισχύουν, πώς αυτό, το 6,8 δηλαδή, συνδέεται στην προσπάθεια να ολοκληρωθεί αυτό το παρόν ε, δημοσιονομικό πλαίσιο και πώς συνδέεται με το επόμενο πολιετές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο. Γιατί κάποια χρήματα θα πρέπει να καταβληθούν και μετά το 2013 ε, για την συνοχή ή για άλλους τομείς που μπορεί να μην τους γνωρίζω. Ερώτημα λοιπόν. Είδαμε στο τέλος του προηγούμενου έτους μια συμβολή περίπου 3,5% που ήρθε από χώρες που ήξεραν ότι μάλλον θα χάσουν τα χρήματά τους. Οπότε αυτό το ερώτημα πρέπει να το θέσουμε ανοιχτά. Είναι δυνατόν να πούμε ότι αυτή είναι η προθεσμία και αν δεν φτάσετε σε αυτή την προθεσμία δεν θα, καταλάβουμε, δεν θα καταβληθούν τα χρήματα και θα τα χάσετε. Αυτό είναι ένα ερώτημα που δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρο για μένα και ίσως κάποιοι συνάδελφοι να το ε, καταλαβαίνουν καλύτερα πώς συνδέονται αυτές οι πληρωμές ε, με, με την έναξη του επόμενου πολιετούς ε, πλαισίου. Ας μου το πούν. Είναι λοιπόν αυτό ένα ερώτημα που είναι πραγματικά δεν είναι πολύ ξεκάθαρο για μένα και αν μπορεί κάποιο να μου απαντήσει ευχαριστώ να τον ακούσω. Ευχαριστώ. Για το θέμα των ράλς. Ήδη έχουμε συμφωνήσει ότι στις 9 Μαΐου θα γίνει μια τεχνική ομάδα εργασίας. Και στις 13 Μαΐου θα συνεδριάσει η πολιτική ομάδα. μάλιστα ένας φιλελεύθερος, ο Γιάνν Μίλλερ είναι ο πρόεδρος εκείνης της ομάδας, οπότε θα τα συζητήσουμε τότε. George Line, George δεν είναι εδώ. Η Μόνικα. Ε, liebe Kolleginnen και Kollegen, ε, zunächst Πρώτα, πρέπει όντως να προχωρήσουμε στο θέμα των πληρωμών. Αφού εγκρίνουμε υποχρεώσεις, κάποια στιγμή θα μας δώσουν και τον λογαριασμό. Οι χώρες γενναιόδωρα εγκρίνουν υποχρεώσεις και μετά διαμαρτύρονται για το υψηλό ύψος των πληρωμών. Για το ε, μεγάλο ύψος μάλλον των πληρωμών. Ασφαλώς είναι περιπλοκή διαδικασία. Βέβαια, θα συζητηθεί εντατικά και με τις χώρες μέλη. Για το νέο προπολογισμό αυτό που με ενδιαφέρει και έρχομαι λίγο σε αυτά που είπε και ο κύριος Άλβαρο προηγουμένως για τις υποχρώσεις δεν βέβαια δεν πρέπει να φανούμε ιστερικοί κατά πόσον δηλαδή οι υποχρώσεις θα πρέπει να διευρυνθούν αφού ούτως ή άλλως δεν τις προλαβαίνουν οι πληρωμές. Είναι μια δικαιολογημένη ερώτηση και πρέπει να τεθεί. Το δεύτερο είναι να, ρωτηθεί, να, να τεθεί ξανά η ερώτηση κατά πόσον τα κονδύλια δαπανώνται ορθά, με τρόπο βιώσιμο. Και τίθηκε το θέμα της ανταγωνιστικότητας το οποίο το έχουμε γράψει στις ατζέντες μας εδώ και χρόνια και παρόλα αυτά η ανταγωνιστικότητα δεν έχει αυξηθεί ε, με ομοιόμορφο τρόπο σε όλες τις χώρες μέλη. ώστε να οδηγήσει και στην δημιουργία επιχειρήσεων και θέσεων απασχολήσεως. Ώστε σίγουρα θα χρειαστεί να γίνουν, να ληφθούν και άλλα μέτρα, όχι μόνο για την απόδοση, αλλά και για τη βιωσιμότητα και την αποδοτικότητα των, των μέτρων να μην τα λέμε ρόδινα για προγράμματα πολλών εκατομμυρίων και τελικώ στην πραγματικότητα μην γίνεται τίποτα. Και μια ερώτηση προς την Κομισιόν. Έχουμε ένα τομέα που μας έχει προκαλέσει πολύ βαριές οικονομικές ζημίες σε όλες τις χώρες μέλη της Ένωσης. Και αναφέρομαι για το, κυβε... για το ε, ε, έγκλημα στον κυβερνοχώρο που έχει φτάσει σε διψήφιους αριθμούς δισεκατομμυρίων. Ένας που κάνει ε, μια ληστεία τράπεζας και ληστεύει μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, το συζητούν όλες οι τράπεζες, ε, συγγνώμη, όλες, το συζητούν όλες οι εφημερίδες και η κοινή γνώμη για μέρες και εβδομάδες. Όμως όταν κάποιος καταχράται δισεκατομμύρια ευρώ στο διαδίκτυο δεν απασχολεί φαίνεται κανέναν. Να εξοπλίσουμε λοιπόν το Cyber Crime Center ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του και να μην είναι και πάλι ένα ρόδινο συνεφάκι το οποίο ε, εμείς εδώ ωρεοποιούμε στην πραγματικότητα όμως δεν μπορεί να λειτουργήσει λόγω έλλειψης προσωπικού και μέσων. Δηλαδή έχει τον ωραίο τίτλο αλλά δεν μπορεί να δράσει γιατί για παράδειγμα για την παιδική πορνογραφία για όλη την Ευρώπη. Υπάρχουν πέντε αρμόδιοι υπάλληλοι για όλη την Ευρώπη για ένα τόσο σοβαρό θέμα όπως η παιδική πορνογραφία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ενώπιον των διαστάσεων, τη της εγκληματικότητας τι προσπάθεια πρέπει να γίνει και επομένως τι αυξήσεις πρέπει ε, να, προβλεφθούν. Και νομίζω ότι πραγματικά αυτό δεν είναι και το μεγαλύτερο κονδύλιο που θα έπρεπε να μας απασχολήσει. Μάλιστα, σας ευχαριστώ. Η Μαρία. Ευχαριστώ Γιούτα. Λυπάμαι που δεν είναι παρόν ο Επίτροπος γιατί έχει σημασία και η παρέμβαση των σκιωδών των σοσιαλιστών σε σχέση με την κατηγορία 4. Θεωρώ όμως ότι τα, οι αξιωματούχοι της Επιτροπής θα διαβιβάσουν τις ερωτήσεις μου γιατί σε σχέση με την ε, κατηγορία 4 αναρωτιέμαι κατά πόσο ελήφθη υπόψη το μέσον ευελιξίας για την χρηματοδότηση της κατηγορίας 4 και αναρωτιέμαι κατά πόσο για το 2013 λαμβάνει υπόψη το οποίο ε, λαμβάνει υπόψη το γεγονός θα πρέπει να προστρέξουμε στο μέσο ευελιξίας και μας ενδιαφέρει να δούμε κατά πόσο θα υπάρχει πλήρης κάλυψη αυτής της κατηγορίας της 4. Για το 11-13, για αυτή την περίοδο, ε, δόθησαν 270 εκατομμύρια ευρώ για προγράμματα γειτονίας του Νότου, δηλαδή τη Μεσογειακή Λεκάνη, την Αραβική Άνοιξη και ούτω καθεξής. Αυτή η συμπληρωματική χρηματοδότηση αφορά την επανακατανομή των πόρων για το προενταξιακό μέσο και το μέσο σταθερότητας καθώς και ε, γειτονίας. Και δεν ξέρω κατά πόσο λαμβάνεται υπόψη το μέσο γειτονίας ιδιαίτερα ως προς τον Νότο ή λαμβάνεται επαρκώς υπόψη το μέσο σταθερότητας μέσα στα πλαίσια της εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης αυτό το έγγραφο δεν γίνεται καμία αμνία για το μέσον για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, το μέσον εταιρικότητας με το, τις βιομηχανικές χώρες, ε, δηλαδή για τις νέες βιομηχανικές χώρες και το μέσο για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη. Έχουν αποκλειστεί από εδώ, τουλάχιστον από αυτή την κατηγορία, ενώ δεν θα έπρεπε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ίσως να λάβουμε και απαντήσεις αμέσως. Ο νέος συνάδελφός μας, ο κ. Πλέκοβιτς. Κροάτης. Ευχαριστώ πολύ και προφέρατε πολύ σωστά το όνομά μου και σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε τον ε, λόγο για πρώτη φορά ως παρατηρητή από το Κροατικό Κοινοβούλιο εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και κάτω από το φως των σχολείων που έκανε ο ε, Επίτροπος Λεβαντόφσκης στη σημερινή του ε, παρουσίαση του προϋπολογισμού του 2013 είπε με κατανόηση ότι η Κροατία αποτελεί ένα πρόβλημα. Δεν θα το έλεγα, ίσως να μην είναι η λύση για την κρίση στην Ευρώπη, αλλά για μας το έτος 2013 θα είναι πολύ σημαντικό διότι στο πρώτο μέρος αυτού του οικονομικού έτους θα ευεργετηθούμε από κονδύλια της προένταξης και στο δεύτερο μισό μετά από την ολοκλήρωση των διαδικασιών κυρώσεως σε όλες τις ε, χώρες μέλη θα πρέπει από τα μέσα του 2013, από τον Ιούλιο δηλαδή, να είμαστε πλήρες μέλος και θα συμμετέχουμε βέβαια και στον σχεδιασμό του προϋπολογισμού για το επόμενο έτος. Και χαίρομαι που ο προπολογισμό που έχει γίνει αντικείμενο διαπραγμάτευση τα τελευταία δύο χρόνια έχει προσαρτηθεί στον προπολογισμό του 2013, ο προπολογισμό που μα αφορά δηλαδή και που περιλαμβάνει τα συμπεφωνημένα μεταξύ των 27 χώρων μελών και της Κροατίας και σε ό,τι αφορά τις δαπάνες αλλά και σε ό,τι αφορά τα έσοδα διότι υπογραμμίζω ότι η Κροατία θα συνεισφέρει στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό ήδη από το δεύτερο μισό του 2013 με συνεισφορά τάξεως μεγέθους των 230 ε, εκατομμυρίων ευρώ. Και για τις πληρωμές για την προένταξη δείχνει όχι μόνο ότι θα περάσουμε από ένα καθεστώς σε ένα άλλο, αλλά και μια αύξηση της απορροφητικότητας σε όλες τις χώρες του εργαλείου ΕΠΑ. Γιούτα Χάουκ. Ολοκληρώσαμε τον κατάλογο των αγοριτών. Τώρα έχουν βέβαια τεθεί ερωτήσεις. Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί κανείς ότι είναι σε θέση να δώσει απαντήσεις. Θα προσπαθήσω να δώσω απαντήσεις ορισμένες από τις ερωτήσεις που τέθηκαν. Του κύριο Κοντμπάνης σχετικά με το ποιο είναι το μερίδιο των εκκρεμών υποχρεώσεων, των resta liquide. Είναι περίπου τα δύο τρίτα του συνόλου που αφορούν τον τομέα της συνοχής. Και ποιο είναι το ποσοστό αύξησης των πληρωμών για το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο. Ο προϋπολογισμός που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπολογίζει τις ανάγκες, τις ελάχιστες απαιτήσει δηλαδή για το 2013, αν αυτές οι πληρωμές δεν είναι διαθέσιμες στο προϋπολογισμό του 2013, μέρος αυτών των απαιτήσεων θα μεταφερθεί στο επόμενο έτος ή στα επόμενα έτη, αναλόγως του μεγέθους. Για τα χρήματα που υπάρχουν για να πληρώνουμε τους λογαριασμούς που θα μας έρχονται, ε, θα τους μεταφέρουμε, αν δεν έχουμε, στον επόμενο προπολογισμό. Για το τίτλο 4, αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει επί του παρόντος την χρήση του εργαλείου ευκαμψίας, η απάντηση για την ώρα είναι όχι. Μετά από σε βάθος αξιολόγηση των αναγκών και κάτω από το περιθώριο δαπανών του τίτλου 4, που είναι υψηλότερο από ό,τι σχεδιαστεί αρχικά είναι περίπου 390 εκατομμύρια. Αυτό επιτρέπει κάποιο περιθώριο ελιγμών για να ρυθμίσουμε με ακριβέστερο τρόπο, εάν καταστεί απαραίτητο, τις πιστώσεις σε ορισμένα προγράμματα και κυρίως για χώρες της, νοτίως της Μεσογείου και ε, της γειτονίας αυτής και για το όργανο, για το για το μηχανισμό γειτονία. Έχει λάβει υπόψη την ανάγκη η Επιτροπή της αύξησης των κονδυλίων, αλλά οι συνθήκες σε ορισμένες από τις χώρες αυτές είναι τόσο επισφαλής για την ώρα, ώστε δεν υπάρχει δυνατότητα να δεσμευθούν και να εκταμιευθούν τα προβλεπόμενα κονδύλια. Θα χρειαστεί λοιπόν να παρακολουθείτε εξέλιξη των συνθήκων στις χώρες αυτές. Τώρα, για το εργαλείο δημοκρατίας και ανθρώπινων δικαιωμάτων, η πρόταση της Κομισιόν είναι να στεθεροποιηθεί σε επίπεδα του 2012 και το παρόν σχέδιο του προϋπολογισμού του 2013. Τέλος, η αύξηση που προτείνεται για τα κονδύλια προένταξης, που και αυτά αυξάνονται σημαντικά, έχουν σχέση με το γεγονός ότι αυτομάτως εφαρμόζονται οι κανόνες για τις υποχρεώσεις και σε αυτά τα κονδύλια και αναμένεται για το 2013 να υπάρξει κίνητρο να αυξηθεί η εφαρμογή για να μην χαθούν τα κονδύλια. Τέλος, Ε, τελευταίο μέρος της απαντήσεώς μου, πάλι για την συνοχή δηλαδή και ορισμένα ε, ερωτήματα του κ. Γκοντμάνης, αν δηλαδή θα πρέπει αυτόματα να προβλέπονται κάποιες προθεσμίες για τις υποχρώσεις για την συνοχή. Υπάρχουν ορισμένες τέτοιες αυτόματες προθεσμίες, νη συν 2 και νη συν 3 ανάλογα με τις χώρες που λαμβάνουν τα κονδύλια αυτά. Εάν δηλαδή αιτήσει χρηματοδότησης δεν ληφθούν μέσα σε μια διετία ή τριετία μετά την ανάληψη υποχρεώσεως, οι υποχρεώσεις αυτές ακυρώνονται αυτομάτως, άρα χάνονται τα χρήματα. Και αυτό είναι και μέρος του λόγου που προκύπτουν οι δυσχέρειες σε ό,τι αφορά την πρόβλεψη με ακρίβεια των υποχρεώσεων που θα πρέπει να αναλυφθούν για τις δαπάνες της συνοχής διότι επί του παρόντος είναι δύσκολο να γνωρίζει κανείς τι θα γίνει το έτος του 2013, πού θα βρίσκονται δηλαδή οι χώρες μέλη, τι θα μπορούν να, ε, τι αιτήσει χρηματοδοτήσεων θα μπορέσουν να υποβάλουν μέσα στην διετία τριετία, στον ίσιν 2 ή ίσιν 3. Ορισμένες από τις υποχρεώσεις αυτές μπορεί να πληρωθούν και το 2014, αφού θα έχουν γίνει ορισμένοι έλεγχοι, αλλά αυτό είναι ένα στοιχείο αβεβαιότητας. Αν όμως οι αιτήσει δεν ληφθούν, τότε βέβαια, όπως είπα, ακυρώνονται αυτομάτως οι υποχρώσεις. Okay. Um, das waren die... Ωραία. Αυτές είναι οι πρώτες απαντήσεις. Ε, προφανώς όσο περνάει ο καιρό θα έχουμε και άλλα ερωτήματα και θα περιμένουμε και περισσότερες απαντήσεις. Οπότε κλείνουμε τη συζήτηση για τον προπολογισμό 2013 και πάμε προς το παρόν βλέπω μόνο τους δύο συνεισηγητές για τις δαπάνες, για το για τις ίδιες, για τους ίδιους πόρους αλλά θα μπορούσαν να μας πούνε οι δύο τι έγινε χτες στο Συμβούλιο, να μας ενημερώσουν. Δεν έχω ιδέα. Ράιμερ, εσύ θέλεις το λόγο, παρακαλώ. Ε, νομίζω ότι πάντα η ομάδα συνεργάζεται καλά, συνεννοείται. Ε, Ακριβώς ε, το θέμα αυτό συζητάται όμως και σε μια άλλη επιτροπή, οπότε πρέπει να πηγαίνω και να ε, έρχομαι. Τη Δευτέρα το απόγευμα κάναμε την ομάδα επαφής υπό τον πρόεδρο Σούλτς. Μετά ε, ήρθαμε σε επαφή χτες την, με την διαπραγματευτική ομάδα πριν από την συνάντηση του Λουξεμβούργο και συζητήσαμε το θέμα και σήμερα στο μεσημεριανό διάλειμμα κάναμε το debriefing με τον Δανό Πρέσβη. Η της συζήτησης του Γενικού Συμβουλίου, του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων είναι κάποιες σκέψεις και στοιχεία τα οποία ίσως θα μπορούσαν να αποτελέσουν κομμάτι του πακέτου του διαπραγματευτικού. Ξεκινούμε με αυτό που ε, είπαμε στην ομάδα επαφής τη Δευτέρα και στα πλαίσια της, ε, του, της συζήτησης που έγινε με τους τρεις ε, προέδρους χτες. Το θέμα δηλαδή του ότι εδώ η διαδικασία της Λισαβόνας, ό,τι αφορά τη συμφωνία και τη συναπόφαση και τις σχετικές διαδικασίες, θα πρέπει να τηρηθεί αυστηρά. Ε, μετά από τη δική μας παρέμβαση, που ίσως να δημιούργησε κάποια έκπληξη στο Συμβούλιο, τέσσερα πράγματα ξεκαθαρίστηκαν, ότι η Δανέζικη Προεδρία ε, είναι υποχρεωμένη, να, νιώθει υποχρεωμένη να τηρήσει τα όσα ε, προβλέπονται από την διαδικασία για τη συμπερίληψη του Κοινοβουλίου όπως έχουμε ξεκινήσει να την εφαρμόζουμε. Δεύτερον, στο πλαίσιο αυτής της ε, συμφωνίας τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί μέχρι να συμφωνηθούν τα πάντα. Τρίτον, υπάρχει εξασφάλιση ότι η αναγκαιότητα να είμαστε σίγουροι ότι αυτά τα πακέτα, τα διαπραγματευτικά, δεν θα προκαταλαμβάνουν την οποιαδήποτε νομοθετική διαδικασία. Από την, και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη σοβαρά από την πλευρά της Δανέζικης Προεδρίας. Και κάποιες λεπτομέρειες θα επανέλθω. Και τέταρτον, η Δανέζικη Προεδρία στο Συμβούλιο του Ιουνίου δεν θα επιμείνει να υπάρξει συγκεκριμένη θέση για τα αριθμητικά στοιχεία ή για τους ίδιους πόρους. Οι διαπραγματεύσεις θα γίνουν, θα συνεχιστούν με βάση αυτά τα διαπραγματευτικά πακέτα. Επίσης, ως συζητητές, στο briefing, μιλήσαμε για τα όσα μας επέβαλε το Συμβούλιο, για την ε, αγροτική πολιτική, για την συνοχή και είπαμε ότι ε, ωραία, καλά κάνατε και το βάλατε εδώ, αλλά εδώ μιλούμε για το μη συναπόφαση. Και αυτό είναι συναπόφαση και αυτό εμπίπτει στη συναπόφαση. Οπότε πρέπει να δούμε στην περαιτέρω διαδικασία πώς από τη μία θα υπάρξουν διάφορε θέσει, γιατί κανένα ακόμα δεν μπορεί, να, δεν, κανένας δεν μπορεί να απαγορεύσει το Συμβούλιο να σκέφτεται, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να βρεθεί μια απόφαση, να ληφθεί η απόφαση ανάμεσα στι διάφορε απόψει που θα ακουστούν στην όλη διαδικασία διαπραγματεύσεων μεταξύ Κοινοβουλίου και των διαφόρων επιμέρου συμβουλίων. Και πρέπει να δούμε τι γίνεται και με τα όσα θα περιληφθούν στην απόφαση που θα μπορούσε να λάβει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και είπαμε ότι θα μπορούσαμε ίσως να προτείνουμε στις ε, συνεδρίες της Δευτέρας Μαΐου μαζί με το Συμβούλιο και, το, και την Κομισιόν να υπάρξει ένα ψήφισμα έτσι ώστε να υπάρξουν ε, σαφή, να καταγραφούν εκεί σαφώς ε, τα σημεία που μας, που μας ενδιαφέρουν. Θέλουμε να επιταχύνουμε τη διαδικασία και ίσως να χρειαστεί να αλλάξουμε λιγάκι την όλη διαδικασία για να μπορέσουμε ταχύτατα να αντιμετωπίσουμε αυτό το, αυτή τη θεματική ενότητα. Η Προεδρία του Συμβουλίου ήταν σχετικά συντηρητική στις ε, απόψεις της ως προς αυτό, αλλά πιστεύω ότι ε, λόγω ακριβώς και των εξελίξεων θα μπορέσουμε να το περάσουμε. Ε, επίσης να υπάρξει μια δήλωση που θα καταγράφει και τις αμοιβέ υποχρεώσεις σε αυτή την όλη διαδικασία. Έτσι ώστε να μην θεωρεί κανείς ότι υπάρχει διακριτική μεταχείριση, να μην μπορεί κανείς να ξεφύγει. Τώρα, για τις λεπτομέρειες, ε, για, τα διάφορα, για τις διάφορες ακαθόδες ε, ε, συζητήσεις για το για την ε, συνοχή και, τον, και την ε, αγροτική ε, πολιτική. Θα μπορείτε να τις δείτε και στο σχετικό κείμενο. Είναι αρκετά ενδιαφέροντα τα στοιχεία. Μετά, έπρεπε να λάβουμε υπόψη μας και το κάναμε με μεγάλο ενδιαφέρον ότι στα έγγραφα τα προσωρινά πρακτικά αλλά και τις δηλώσεις τύπου υπάρχουν ε, κάποιες, υπάρχει μια διατύπωση την οποία την αναφέραμε και σήμερα ε, λέει, σα παραθέτω ε, στα αγγλικά, η γενική προσέγγιση είναι μια πολιτική συμφωνία του Συμβουλίου με, την, ε, ε, αναμένοντας να υιοθετηθεί η πρώτη θέση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όσο εδώ καλά, η γενική προσέγγιση για, το νομοθετικό πακέτο για την πολιτική συνοχή είναι μερική, είναι, δεν είναι πλήρης, γιατί κάποια, κάποια στοιχεία εξαιρούνται και πρέπει να δούμε το θέμα τη επληξιμότητα κάποιων περιφερειών τα οποία θα, οι οποίε θα συμφωνηθούν στα πλαίσια του νέου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Τελεία. Είχαμε πει ότι το κείμενο αυτό βεβαίως είναι ευθύνη των υπηρεσιών του τύπου και δεν νομίζω ότι μια τέτοια έκφραση θα έπρεπε να περιλαμβάνεται εντάξει, δεν φταίνε οι διερμηνεί. γι' αυτό προφανώ φταίει ο τύπο. Το γραφείο τύπου. Ε, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του ε, Δεκεμβρίου του 2005 από την ε, σελίδα 5 ως το 25 περιλαμβάνουν πολλά μικρά αριθμητικά στοιχεία, ποσοστίας, μονάδες κτλ. που τότε μπορεί να ήταν επιθανές ή προφανείς, αλλά που δεν θα έπρεπε να βρίσκονται μέσα στην απόφαση. Γι' αυτό λοιπόν αυτό είναι σημαντικό να το έχουμε υπόψη μας. Γι' αυτό το συζητήσαμε και το τονίσαμε ιδιαίτερα. Και τα, οι ίδιοι πόροι είπαμε ότι θα μπουν στα τέλη Μαΐου στην προετοιμασία που θα γίνει για το σχετικό δημοσιονομικό ε, ε, πακέτο διαπραγμάτευσης. Συγγνώμη. Πρέπει λοιπόν όλα αυτά να ληφθούν υπόψη γιατί ε, πρέπει να υπάρχει συνέπεια μεταξύ των ιδιών πόρων, των αριθμητικών στοιχείων του πολιετούς πλαισίου και της ευελιξίας που πρέπει να έχουμε για την προετοιμασία ε, που θα κάνει και η ε, Προεδρία. Αυτά από μένα. Ζητώ συγγνώμη. Αλλά έχουμε συμφωνήσει μεταξύ μας τόσο καλά που αν ακόμη και αν λείπω εγώ, ο συνάδελφος θα πει περίπου τα ίδια. Ωραία. Υπάρχουν ερωτήματα. Αν υπάρχουν, θα τα απαντήσει ο συνάδελφος. Δεν υπάρχουν. Ωραία. Προσθήκες δεν υπάρχουν, επιπλέον σχόλια όχι. Πολύ ωραία. Πάμε τώρα στο σημείο 6. Α, όχι, όχι. Αναβάλλετε το 6 γιατί η Φραντσέσκα Βαλζάνη δεν είναι εδώ. Πάμε στο 8. Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κοινωνική αλλαγή και την κοινοτομία. Η Εστέλ κάνει την, εκπονεί την νομοδότηση αυτή. Να της δώσουμε το λόγο. Oui, merci, Madame Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να σας υπενθυμίσω ότι το πρόγραμμα για την κοινωνική αλλαγή και την καινοτομία είναι μια πρόταση επιτροπής για την ομαδοποίηση τριών μέσων που ήδη προϋπάρχουν, πρόγρας, έρες και το Ευρωπαϊκό Μέσο Μικροχρηματοδότησης, Progress για ε, λόγους απλούστευσης ήδη κατά μια προγενέστερη ανταλλαγή απόψεων είπε ότι η ομαδοποίηση ε, οδηγεί σε ορισμένα ζητήματα έτσι ώστε να δούμε τη στοχοθέτηση, τους δικαιούχους και τα μέσα. Και δεν θα πρέπει παρά να υπάρχει συνοχή, δεν πρέπει να την χάσουμε. Ως προς προτάσεις που διατύπωσα για να ε, βελτιώσουμε το πλαίσιο, θα ήθελα να πω ότι σε αντίθεση με αυτά που είπε η Επιτροπή ότι δεν πρέπει να κρίνουμε τα μέσα, τους ανάλογα με το, τα, τα μέσα ανάλογα με το μέγεθός τους αλλά με την προσθέμενη αξία το είδαμε με ορισμένα μικροσχέδια σε ευρωπαϊκό επίπεδο στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Μικροχρηματοδότησης. Ως προς το Μηχανισμό Μικροχρηματοδότησης θα πρέπει να προωθηθεί και αναφέρουμε ότι αν η πρόταση της Επιτροπής επιτρέψει να εξασφαλίσουμε στο μηχανισμό χρηματοδότησης, ξεχνά έναν επιπρόσθετο μηχανισμό, δηλαδή τα συνοδευτικά μέτρα για ένα μέρος του κοινού και θεωρούμε ότι θα πρέπει να αναζητηθεί αυτός ο συμπληρωματικός χαρακτήρας με συνοδευτικά μέτρα από το ΕΚΤ σε δημοσιονομικά πλαίσια και με την εισηγήτρια και τους σκιώδεις προτείνουμε μία κλίδα κατανομής ε, των προγραμμάτων διαφορετική από αυτή που προβάλλει η Επιτροπή και θεωρούμε ότι ως προς τα διοικητικά έξοδα της Επιτροπής θεωρούμε ότι θα πρέπει να ανέλθουν αυτά τα έξοδα στο 2%. για τις διοικητικές δαπάνες. Φαίνεται ε, ότι σε δημοσιονομικό επίπεδο μας ενδιαφέρει η ε, σταθερότητα και γι' αυτό αποφασίσαμε να αναβάλουμε την έγκριση των ποσών περιμένοντας το πολιετές ε, πλαίσιο και, θα το, και σε σχέση με τον Ιούνιο του 2011 έχουμε μια αύξηση της τάξης του 5% για τον προϋπολογισμό του 2013. Αυτά ήθελα να σας πω συνοπτικά, Πρόεδρε. Για την τροπολογία η προθεσμή είναι αύριο στις 10 και θα εγκριθεί στις 31 Μαΐου από την Επιτροπή μας η έκθεση αυτή. Ich habe jetzt nur eine Wortmeldung. Ένα ζητάει μόνο το λόγο, κύριος Γιακοσλόφσκι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Γκρελιέ για την έκθεσή της και για τα σχόλια. Θεωρώ ότι θα πρέπει να έχουμε ένα ενιαίο πρόγραμμα. Πράγματι, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα προς τον συντονισμό των δράσεων στον τομέα της απασχόλησης και της κοινωνικής ε, πολιτικής και για την ευθυγράμμιση των διαδικασιών. Συμφωνώ με την εισηγήτρια ότι για την κοινωνική καινοτομία θα πρέπει να υποστηρίξουμε όχι μόνο τα μεγάλα αλλά και τα μικρομεσαία ε, σχέδια και προγράμματα θα πρέπει να ε, δοκιμάσουμε νέες λύσεις σε όχι τόσο υψηλή κλίμακα. Θα πρέπει να δούμε κατά πόσο μπορούμε να επιτύχουμε μια ε, να φτάσουμε σε μια κρίσιμη μάζα χρηματοδοτώντας μεγάλα σχέδια. Αυτό λεγόταν μέχρι τώρα, αλλά νομίζω ότι δεν είναι σωστό. Σε σχέση με την οργάνωση διασκέψεων, συμφωνώ με τα σχόλια της κυρίας Γκρελιέ, θεωρώ ότι η χρηματοδότησή τους για τον κοινωνικό αποκλεισμό, την καταπολέμηση της φτώχειας και συναφή θέματα συμβαδίζει με τους στόχους αυτού του προγράμματος και γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να ε, υπάρχει αυτή η δυνατότητα, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι οι διασκέψεις θα πρέπει να υπόκεινται στους στόχους του προγράμματος. Επίσης γίνεται λόγος για μια νέα κατανομή ανάλογα με τα τμήματα του προγράμματος Αναρωτιέμαι κατά πόσο δεν θα έπρεπε να αρκεστούμε στην ε, πρόταση επιτροπής, δηλαδή οι αλλαγές ε, βρίσκονται πέραν, ε, κινούνται πέραν από τις δικές μας αρμοδιότητες. Δεν μπορούμε να μειώσουμε τις δαπάνες του προγράμματος Progress, το Eures, είναι εντελώς νέο και διαφορετικό από ό,τι γνωρίσαμε μέχρι τώρα. Νομίζω ότι ο διαχωρισμός μεταξύ των διαφόρων τμήματων, η κατανομή κονδυλίων θα πρέπει να αναθεωρηθεί. Συμφωνώ με την προσέγγιση της Επιτροπής, αλλά προτείνω και μία άλλη λύση, δηλαδή ε, να έχει η Επιτροπή διακριτική ευχέρεια στην χρηματοδότηση των διαφόρων προγραμμάτων και στη μεταφορά πόρων μεταξύ των διαφόρων προγραμμάτων μέχρι ένα 5%. Βεβαίως η αρμόδια του προϋπολογισμού αρχή θα ενημερωθεί για αυτές τις ενδυνάμει μεταφορές. Και πιστεύω επίσης ότι θα πρέπει να συντονίσουμε το συμπληρωματικό χαρακτήρα και την αποδοτικότητα αυτών των προγραμμάτων. Ja, vielen Dank. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ. Αύριο το μεσημέρι λίγου ή λίγη η προθεσμία κατάθεση των τροπολογιών. Η ψηφοφορία θα γίνει στις 31 Μαΐου. Εστέλ, παρακαλώ να απαντήσω στο συνάδελφο για την κατανομή μεταξύ των διαφόρων προγραμμάτων. Το είδαμε με, μαζί με τους εκπροσώπους της Επιτροπής Απασχόλησης και άλλους συνεισηγητές για να υπάρξει μεγαλύτερη ελαστικότητα. Θα πούμε ότι αυτό θα είναι ε, ενδεικτικό για να ε, ε, αντιμετωπίσω και μετριάσω την ανησυχία σας. Είναι ούτως ή άλλως ενδεικτική μου, μου πληροφορούν. Καλά λοιπόν, ευχαριστώ πολύ λέει η Γιούτα Χάουκ. Αν άλλος κανείς δεν επιθυμεί να ε, λάβει το λόγο, τότε θα αναμένουμε τις τροπολογίες που θα υποβάλουν οι συνάδελφοι, με σίγουροι, κατά Και ας έρθουμε τώρα στο 9. Το πρόγραμμα δράσης για την υγεία. Η κυρία Βέρτμαν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. 10 περίπου της 100 του ΑΕΠ απορροφά αυτός ο κλάδος της υγείας δηλαδή. Είναι πιο τους σημαντικούς. Και εκεί μάλιστα απασχολείται και το δέκατο όλων των απασχολουμένων. Αυτά σημαίνουν περισσότερη ποιότητα ζωής και ένα σημαντικό κινητήρα ανάπτυξης για τις κοινωνίες μας, ιδίως μέσα στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης. Προτείνει τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το τρίτο πρόγραμμα δράση. Υγεία για την ανάπτυξη μέσα στα πλαίσια του επόμενου πολιετού δημοσιονομικού προγράμματο με τέσσερι επιμέρου στόχου και με σημαντικό δυναμικό ανάπτυξη. Αφενό καινοτόμα και βιώσιμα συστήματα υγεία, Δεύτερο, περισσότερη πρόσβαση σε καλύτερε και ασφαλέστερες υπηρεσίε υγεία, Τρίτο, πρόληψη ασθενειών και προώθηση της υγείας. Και τέλος, προστασία των πολιτών απέναντι σε ε, ε, ε, απειλές της υγείας που διαβαίνουν τα σύνορα. Αυτά για μέχρι το 2020 βλέπουμε ότι λείπει περίπου ένα εκατομμύριο απασχολούμενων στον τομέα της υγείας. Και αυτή η ανάπτυξη του τομέα υγείας θα δώσει και μια δυναμική και στην απασχόληση. Προτείνει λοιπόν 466 εκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2020 60% των χωρών μελών για... και μπορεί να φτάσει και μέχρι 80% η συγχρηματοδότηση. Οι τροπολογίες που προτείνω εγώ αναφέρονται στα πιο σημαντικά που γίνονται ορισμένε προβλέπω ορισμένε συμπληρώσει και στα σημεία όπου μου φαίνεται το κείμενο τη Κομισιόν να δίνει αφορμή σε παρανοήσει ή είναι κάπω αδύναμο, και θα παρακαλέσω όλες και όλους τους συναδέλφους αν έχουν άλλες ιδέες να συζητήσουν μαζί μου, να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις διατυπώσεις και πολύ θα χαρώ να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε και σε συμβαστικές τροπολογίες. Το συμπέρασμα είναι ότι πρέπει να δούμε μακροπρόθεσμα τι γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μειώνεται ο πληθυσμός της Ευρωπαϊκής Υπήρου και μειώνεται η αριθμή μας και γερνάμε. Αν θέλουμε να διατηρήσουμε την ανταγωνιστικότητά μας λοιπόν πρέπει να αρχίσουμε να δραστηριοποιούμαστε εδώ και τώρα και όχι σε 10-20 χρόνια. Και αυτό το θέμα της υγείας και από οικονομική άποψη έχει πολύ μεγάλη σημασία. Εγώ θεωρώ ότι η Κομισιόν δρά ορθά και θα πρέπει να υποστηριχθεί η πρότασή της στο κατάλληλο πλαίσιο. Οι τροπολογίες αναμένονται μέχρι τις 7 Μαΐου. Η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας προβλέπεται για την 31η Μαΐου. Αναμένω με μεγάλη ανυπομονησία και ενδιαφέρον τις συζητήσεις. Κοιτάξτε τώρα, εγώ είμαι και σκιώδης εισηγήτρια για τη γνωμοδότησή σας, λέει η κυρία Χαουκ. Οι τροπολογίες που άπτονται του προπολογισμού μου φαίνονται σωστές και τις υποστηρίζω όλες. Φαντάζομαι θα τις έχουν δει και οι συναδελφοί μας και μιλώ για τις 1, 2, 4, 7, 12 και 14 που νομίζω ότι είναι εντάξει. Αναφέρονται πράγματι στα δικά μας καθηγόντα στις δικές μας αρμοδιότητες. Οι 3, 5, 6, 9 και 15 αυτές άπτονται μάλλον της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Κατ' ουσίαν, δηλαδή, σε ό,τι αφορά το σιώδες περιεχόμενό τους, ε, αν πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές. Πιστεύω πάντως, κυρία Βέρτμαν, κυρία Βέρτμαν, ότι εν πάση περιπτώσει... Καμιά φορά βέβαια επικαλύπτονται οι τροπολογίες, αλλά τέλος πάντων η τροπολογία που διευρύνει το πεδίο εφαρμογής, όχι δηλαδή μόνο για την κατάχρηση των ενοπνευματοδών και του καπνού, αλλά και των ναρκωτικών και τις σχετικές συνέπειες, εκεί θεωρώ ότι εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είμαστε διόλου σε θέση να κάνουμε τίποτα. Γιατί αυτό ξεφεύγει απολύτως από την αρμοδιότητά μας. Η κατάχρηση ναρκωτικών για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ζήτημα ποινικού δικαίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καμία σχέση με το ποινικό δίκαιο. Στη χώρα μου στη Γερμανία το, ο νόμος περί ναρκωτικών λέει βέβαια ότι απαγορεύεται η χρήση καταρχήν ναρκωτικών ουσιών αλλά δεν διώκεται αυτός που ποιείται προσωπική χρήση. Παρ' όλα αυτά δεν μπορούμε να αγγίξουμε αυτή την πρόληψη. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι με τον οργανισμό που έχει την έδρα του στη Λισαβόνα να παρακολουθήσουμε τους δρόμους που παίρνουν τα παράγωμα ναρκωτικά και να προσπαθήσουμε τέλο πάντων να βρούμε από πού διαβαίνουν αυτά και σε συνεργασία με τρίτες χώρες να κλείσουμε τις διόδους αυτές. Κατά τα άλλα τα χέρια μας είναι δεμένα. Για καπνό και ε, ενόπνευμα, εκεί αυτά είναι νόμιμα εντός εισαγωγικών ναρκωτικά. Αυτά εντάσσονται βέβαια στο πρόγραμμα δράσης για την υγεία και πάντοτε έχουμε κάνει σχετικά, σχετικές δράσεις. Το πρόγραμμα δράσης για 7 χρόνια προβλέπει λίγο πάνω από 400 εκατομμύρια ευρώ. Ούτω ή άλλω δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν τα πάντα που ίσω θα ήταν αναγκαία για την προστασία τη δημόσια υγεία. Αλλά να προωθηθούν κάποια παραδείγματα καλών πρακτικών, αυτό είναι ίσω δυνατό και σκόπιμο. και για την ε, υποχρέωση υποβολής ε, αναφορών και για τα κριτήρια που θα πρέπει τα ε, κριτήρια αξιολόγησης να είναι από πριν καθορισμένα. Εγώ βρίσκω ότι είναι σωστό αυτό και είναι άλλωστε και δικής μας αρμοδιότητας ως Επιτροπής Προϋπολογισμών αφού στο κάτω της γραφής εμείς είμαστε υπεύθυνε για να δούμε να χρησιμοποιούνται σωστά τα σχετικά κονδύλια. Μάλιστα, λοιπόν, τώρα ξαναγίνομαι προεδρεύουσα τη Επιτροπή Προπολογισμών. Άλλο κανεί. Α, ναι, η κυρία Μαζόνη. Εγώ είμαι σκιωδής από το ΕΛΚ. Νομίζω ότι η πρόταση της Επιτροπής μας βρίσκει σύμφωνους διότι εναρμονίζει το πρόγραμμα για την υγεία με τους στόχους της Στρατηγής Ευρώπη 2020 και βασίζεται σε ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να προωθήσει την καινοτομία και την βιωσιμότητα καθώς και την συμμετοχή. Μιλάμε για καινοτόμες λύσεις έτσι ώστε να φτάσουν σε αποτελεσματικότητα, να αντιμετωπίσουμε την έλλειψη προσωπικού και να τοποκριθούμε στις ανάγκες του πολίτη. Το σημείο εκκίνησης αφορά την υγεία ως ε, παράγοντα ανάπτυξης και μας ενδιαφέρει η επίπτωση της υγείας των πολιτών για την ανάπτυξη της οικονομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρώ ότι μπορώ να συμμεριστώ την παρατήρηση της εισηγήτριας σε σχέση με τα επιπρόσθετα πόσα, έτσι ώστε να δούμε την επίπτωση αυτού του τομέα στο διορθωτικό προϋπολογισμό. Θα πρέπει λοιπόν να ξαναδούμε τις πιστώσεις, αλλά δεν έχω εγώ αρμοδιότητα για κάτι τέτοιο. Συμμερίζομαι και τις προτάσεις της εισηγήτριας αλλά θεωρώ ότι η συγγήτρια στέκεται στο να υπογραμμίσει την ανάγκη να δράσουμε στον τομέα της πρόληψης ε, καταπολεμώντας τη χρήση του αλκοόλ και την καταπολέμηση της χρήσης των ναρκωτικών. Γίνεται λόγος και αναφορά στα ναρκωτικά και η συγγήτρια ζητά μία τροποποίηση έτσι ώστε να λάβουμε υπόψη και το κριτήριο της παχυσαρκίας για να δούμε ποιοι είναι και οι παράγοντες ε, διατροφής που υπησέρχονται. Αυτό μπορούμε να το συμμεριστούμε. Όμως δεν μπορούμε να δεχτούμε την καταπολέμηση χρήσης καπνού και αλκοόλ, διότι η Κομισιόν απαριθμεί τους παράγοντες σαν να πρόκειται για μία ε, ιεράρχηση, στενή ιεράρχηση των κινδύνων και του πρόωρου θανάτου. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανισορροπία σε μεγαλύτερες ανισορροπίες ως προς την κατανομή και απόδοση ευθυνών και θα πρέπει να δούμε και άλλους παράγοντες κινδύνου που, αφορά τη μόλυνση έθνης, που αφορούν τη μόλυνση του περιβάλλοντος και ούτω καθεξής. Θα πρέπει να οριστεί ένας απογραφικός κατάλογος ο οποίος να είναι χρήσιμος για την πλήρη πρόληψη και θα πρέπει να μιλήσουμε και για χρόνιες ε, και για χρόνιες ε, παθολογίες που αφορούν τη μόλις του περιβάλλοντος, τα νόξ και ούτω καθεξής, διοξίδιο του άνθρακα κλπ. Και την έλλειψη φυσικής δραστηριότητας, γιατί και αυτό αυτό υπησέρχεται στους παράγοντες όπως μας δείχνουν πολλές μελέτες που έχουν αναλυφθεί από τον ΠΟΗ. Αυτή είναι μία, αυτή είναι μία από τις βασικές αιτίες το, της, ε, των χρονίων ε, παθονοσημάτων, παθολογικών νοσημάτων. Νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να βελτιώσουμε το κείμενο Και ως προς παράγραφο 6, καλούμε τα κράτη-μέλη να εντάξουν τα εθνικά προγράμματα την υγεία ως προτεραιότητα με βάση τους πόρους που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η ένδειξη, αυτή η μνήα δεν αντικατοπτρίζεται αργότερα στις ρυθμίσεις. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να ε, της δοθεί και μία συνέχεια ε, ως και να θεωρηθεί κριτήριο επιλεξιμότητας. Στην παράγραφο 10 γίνεται λόγος για κάποια προτίμηση για χώρες που έχουν ε, ε, ΑΕΠ κάτω από 90% για να προωθήσουμε την υγεία. Νομίζω ότι δεν πρέπει να ληφθεί υπόψη αυτή η διαφοροποίηση, να υπάρχουν ίση όροι πρόσβαση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος, στην παράγραφο 16 γίνεται λόγος για κριτήρια επιλεξιμότητας, αλλά το θέμα δεν εμβαθύνεται στη συνέχεια. Θα πρέπει λοιπόν στον ίδιο τον κανονισμό να γίνει λόγος για το ε, κριτήριο πολλαπλών κονδυλίων ή ταμείων και η παράγραφος 20 αναφέρεται στη διαχείριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι η διατύπωση δεν λαμβάνει υπόψη την ε, διαστρωματική διακυβέρνηση που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη σε όλες τις δραστηριότητες που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές είναι οι υποδείξεις μου προς την εισηγήτρια. Ευχαριστώ. Ja, vielen Dank. Ähm, Ευχαριστώ. Μπορώ να υποστηρίξω σε πολλά σημεία αυτά που λέτε. Αλλά εφόσον δεν μιλούμε για θέματα προπολογισμού, τις τροπολογίες μας θα πρέπει να τις ε, υποβάλλουμε στην Φρανσουάς ε, Γκροστέτ που είναι η υπεύθυνη για, από την Επιτροπή ε, Περιβάλλοντος. Όλα λοιπόν όσα θέλουμε να αλλάξουμε στο κείμενο της Κομισιόν ουσιαστικά θέλουμε να αλλάξουμε όχι τα νούμερα, όχι δηλώσεις αλλά για την εφαρμογή αυτά θα πρέπει να τα στείλουμε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Δεν μπορούμε να κάνουμε εμεί την πολιτική για την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Εμείς κάνουμε την γνωμοδότησή μας που θα ασχοληθεί με το τι θα κάνουμε με τον προπολογισμό. Απλώς για να τα ξεκαθαρίζουμε λιγάκι. Άλλος κανείς. Κυρία Βέρτμαν, θέλετε να κλείσετε. Να ευχαριστήσω τη συνάδελφα για τις παρατηρήσεις. Μπορούμε να κάτσουμε και δυο μαζί και να βελτιώσουμε το κείμενο που χρειάζεται. Ευχαριστώ. Ωραία. Άρα τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Στο... Φτάσαμε στο τέλος της ημερήσιας διάταξης. Δεν φτάσαμε στο τέλος μας, φτάσαμε στο τέλος της ημερήσιας διάταξης. Ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους που Έφτασαν μέχρι αυτή την ώρα που έμειναν εδώ. Η επόμενη συνεδρίασή μας είναι στις 8 Μαΐου. Θα τα πούμε λοιπόν στις 8 Μαΐου στις 3 το μεσημέρι. Ως τότε, καλό απόγευμα.